Συνάδελφοι, λέει η Πρόεδρος. Γύρισαμε από τις ε, διακοπές και ανταλλάσσουμε εντυπώσεις. Ξέρω ότι έχετε υποχρεώσει άλλες επιτροπές και θέλετε να προχωρήσουμε προς την ψηφορία. Οπότε ας ξεκινήσουμε την ημερήσια διάθεση. Οπότε ε, καλώς ορίσατε πρώτα-πρώτα, ήρθατε στην ώρα σας. Αυτό είναι καλό για την καινούργια χρονιά. Είμαστε όλοι επιμελείς μαθητές και ήρθαμε για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ελπίζω ότι πέρασε καλά στις διακοπές. Είχαμε ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι στη χώρα μας. Έλλειψη βροχής, πολύ ζέστη. Ε, ευχάριστα πράγματα. Για να δούμε τώρα. Ημερήσια διάταξη. Πρώτα-πρώτα. Χτες πήρατε το email που λέει ότι έχουμε προσθέσει δύο θέματα. Τρία. Στην μέσα διάταξη θα τα συζητήσουμε αύριο. Πρώτα πρώτα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες για την διάσκεψη για το κλίμα. COP24 του Πόσνα νομίζω. Δεν είμαι τόσο σίγουρος αν πρόκειται για το Πόσνα. Τέλος πάντων. Έχουν πάντα τις σχετικές τροπολογίες για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που θα αφορά την ε, ΚΟΠ, τις συνομιλίες για το κλίμα. Αυτό θα είναι το θέμα 18. Άλλα δύο θέματα μετά για τα ανθρωπιστικά. Είχαμε κάποιες ε, εξελίξεις ε, ανησυχητικές. Θα είναι το θέμα 19 όσον αφορά την λόριδα της Γάζας. Και κατόπιν το 20 για την Βενεζουέλα. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά έχουν μεταβεί εκεί. Και να συζητήσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Ε, τα ακούσαμε και στο BBC και για τις δύο αυτές ε, περιοχές, Γάζα και Βενεζουέλα. Αυτά για αύριο το πρωί. Και να δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Πρώτη ενημέρωση. Επομένως συμφωνείτε με αυτή την τροποποίηση μες διάταξης. Ωραία. Ανακοινώσει της Προέδρου που είναι το δεύτερο θέμα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την ετήσια συνάντηση μεταξύ Ευρωβουλευτών και επικεφαλής των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Αυτό θα γίνει το απόγευμα. για την ανταπόκριση, την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις παγκόσμιες προκλήσεις, ε, μετανάστευση, χαίρετε έχουμε πολλές, πολλούς φορείς ε, που ασχολούνται με αυτά. Έχουμε για τους βιώσιμους στόχους την διάσκεψη της ε, Νέας Υόρκης που έγινε λίγο πριν τις τέρνες διακοπές και τελικά δεν προσυπέραψαν οι Αμερικανοί την τελική διάσκεψη και βλέπουμε ότι οι πολυμερείς οργανώσεις, φορείς, οργανισμοί βρίσκονται τώρα υπό πίεση αυτά, θα συζητήσουμε. Επίσης θα συμπροεδρεύσουμε τον Κλοντ Μωράες της ΛΥΜΠΕ για μια συνάντηση που έχει τον τίτλο «Διαχείριση της μετανάστευσης» στα πλαίσια του Συμφώνου του ΟΗΕ το 3G3 μεταξύ 4 παρατέταρτο και 5 και 4 την Τρίτη την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για να γραφτείτε για τις διάφορες επιμέρους συναντήσεις αυτής της εκδήλωσης Τέλος πάντων θα ενημερωθείτε και αν θέλετε να πάτε να το πείτε. Τους ξέρετε αυτούς τους πρεσβευτές μας, τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Ε, είναι ενδιαφέρουσες συναντήσεις μαζί τους και θα είναι ενημερωτικές. Επίσης, έχουμε τις αποφάσεις των συντονιστών, η συνάντηση της 11ης Ιουλίου, έχετε λάβει τα σχετικά. Εάν δεν υπάρξει κάποια ένσταση, θα θεωρηθεί ότι τα εγκρίνεται. τεσσερα Έγκριση πρακτικών 16η-17η Μαου, 25 Ιουνίου. Τα έχετε λάβει και εδώ πάλι μέχρι το τέλος της συνεδρίας, αν δεν έχουμε ενστάσεις, θεωρούνται τα πρακτικά έγκριθέντα 5. Καλώς ορίσατε συνάδελφοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχετε κάποια ανακοίνωση. Όχι. Ε, διακοπές ήταν. Καλά, όσο προχωράει η χρονιά θα προκύψουν οι ανακοινώσεις. Άρα, πάμε στις ψηφοφορίες. της κάρτας σας βάλτε στο μηχάνημα. Έχουμε δύο θέματα προς ψήφιση. Το πρώτο, το έξι τη θάσευση παγκοσμιοποίησης εμπορικές πτυχές. Πρέντα είναι ο εισηγητής μας, ο οποίος απουσιάζει. Δεν υπάρχει κάτι από πλευράς του, άρα το ψηφίζουμε. 6. Τη θάσευση παγκοσμιοποίησης. Έχουμε κάποιες συμβαστικές και ξεκινούμε με την υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη συμβαστική 2 ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική. τρία, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έντεκα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, και καταπίπτει το δεύτερο τμήμα, δεν θα έπρεπε να γίνει, πρέπει να γίνει ψήφιση. 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παραλείψαμε Κάποια ψηφοφορία. Μετά το 10. Α, πρέπει συνεργαθεί. Και ε, κοιτάξτε την πρώτη σελίδα της λίστας. Θα έπρεπε να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα του 10. Θα έπρεπε να ψηφιστεί. Εγώ φταίω. Δεύτερο τμήμα του 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε. Συμβαστική 5. Στην τρίτη σελίδα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική παριθμών 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι επόμενες καταπίπτουν και πάμε στο συμβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για το 38. Πέρασε. Απορρίπτεται. 39 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του 39 ψηφίζουμε νομίζω εγκρίνεται ψήφισαν όλοι πέρας εγκρίνεται όντως 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 8. Βλέπετε που είναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας. εγκρίνεται οριακά. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για το 51. Πέρας. Εγκρίνεται. 52 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πενήντα έξι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, όχι, όχι. Έχετε δίκιο. Πρώτα την συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 9 και τώρα πάμε στο 56 δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα του 56 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του 56 ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 61 πέρας εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 62 πέρας εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε ψηφίζουμε Πέρας. Έγινε με ευρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Πρέντα που είναι απόν. Φαντάζομαι ότι θα του το διαβιβάσετε και σας ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε. Προϋπολογισμός. Δύο τμήματα. Έχουμε δύο διαφορετικές λίστες για ψηφοφορία. Πρώτα-πρώτα τις ε, τροπολογίες και κατόπιν το ψήφισμα. Ξεκινούμε με τις τροπολογίες. Άρνε Λίτς. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ε, πως ε, και ελπίζω μάλιστα το καλοκαίρι ήταν καλό για όλους. Είχαμε πολλές ε, θετικές εξελίξεις στα διεθνή φόρα, η συνεισφορά λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε αισθητή, συζητήθηκε η διπλωματία για το κλίμα και δείξαμε ισχυρή παρουσία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους για την ιδιαίτερα καλή συνεργασία στις ε, τροπολογίες του προπολογισμού και μάλιστα μια συνεργασία που ήταν ιδιαίτερα καλή δεδομένων των θερινών διακοπών. Συζητήθηκε η ανθρωπιστική βοήθεια, η Τουρκία, ε, ανταλλάξαμε email με τους κοιόδης εισηγητές για την ανάγκη να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ε, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, να μην κλείσουν πόρτες. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους και ε, ανυπομονώ για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Πολύ ωραία, μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Αρχίζουμε με τις τροπολογίες και θα σας διαβάσω τα νούμερα. 55-62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55-52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55-53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55-56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55-57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55-66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55-78 υπέρ κατά, αποχές, 5561 55-61 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 5561 61 Τροπολογίες από Γκερέρο, Φρουντζούλιτσα, Νόιχλ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται 5563 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55-59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55-65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55-76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55-60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55-68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55-58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55, 77. εβδομήντα εφτά υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε γιατί νομίζω πως υπάρχει μια, ένα μπέρδεμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται μάλλον. Πέρας. Ναι, ναι, απορρίπτεται. 55-64. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55-75. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. του κυρίου Πεϊόν. Υπέρ. Μάλιστα, ε, διαφωνείτε με την προφορική τροπολογία, δεν μπορούμε λοιπόν να την ψηφίσουμε. Περνάμε στην 5550. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 5573. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5574. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5572. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5570. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5569. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5551. Υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 5551. Πέρας. Εγκρίνεται. 5567 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτά για τις τροπολογίες. Περνάμε λοιπόν στο ψήφισμα.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 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος στην 11. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. έλεγχο στη 13. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 15. Ψηφίσατε. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά.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 Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 28. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Θέλετε να πείτε κάτι? Δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι έγινε ένα λάθος στην 16. 17. Λάθος ψήφισα. Μπορούμε λοιπόν να το διορθώσουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε την ε, ψήφο. Όχι, όχι, λυπάμαι τελείωσε η ψηφοφορία. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει μηχανισμός διόρθωσης στην Επιτροπή. Μπορείτε να βάλετε κάποια υποσημείωση για την Ολομέλεια. Είναι εξάλλου γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προπολογισμών. Εμείς όμως δεν μπορούμε να αλλάξουμε αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. 30 του κυρίου Ρούμπιγκ. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Χάνεις και κερδίζεις. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε την 31.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 Πέρας. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 43. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές ελέγχουμε τη 48. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης με ονομαστική κλίση όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστούμε πολύ, Άρνα. Και σας ευχαριστώ όλους. Εδώ φτάσαμε στο τέλος των ψηφοφοριών για σήμερα το πρωί. Καλώ συνάδελφοι. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα, παρακαλώ να το κάνουν για να προχωρήσουμε στο σημείο 8. Αθέμητες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Παρακαλώ, εάν θέλετε να Αποχωρήστε από την αίθουσα, εκεί μπορείτε να βγείτε από την αίθουσα και να συνεχίσετε να φλιαρείτε, να μιλάτε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Τώρα όμως εδώ ε, θα εξετάσουμε το ε, σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Άγκρη. Περί πρόκειται. Στις να σας κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις πρώτα και μετά θα προχωρήσω στις δικές μου τροπολογίες. Στις 12 Απριλίου η Επιτροπή πρότεινε οδηγία για θέμητες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων και η ιδέα είναι να απαγορευθούν οι πιο επιβλαβείς και καταστροφικές αθέμητες εμπορικές πρακτικές για να προστατευτούν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί. Όλοι ξέρετε περί πρόκειται είναι παράπονο των αγροτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός, ε, έτοιμα για πάρα πολλά χρόνια, ότι δηλαδή τα μεγάλα ε, σούπερ μάρκετ τους ασκούν τεράστιες πιέσεις για να μειώνουν τις τιμές τους χρεώνουν για να μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα στις προθήκες των σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Είναι πολύ μακριά η διαμάχη αυτή ε, για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ορισμένες χώρες ήδη έχουν υιοθετήσει νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο για να προστατεύσουν τους αγρότες και τους παραγωγούς και χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια και αυτό προσπαθεί η Κομισιόν να κάνει με την ανάληψη πρωτοβουλία για αυτή την οδηγία και οι ευρωβουλευτές το ζητούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα τα ψηφίσουμε όλα αυτά ε, στις αρχές Οκτωβρίου. Γιατί κάνουμε εμείς γνωμοδότηση, συντάσσουμε ως ΝΤΕΒΕ, ως Επιτροπή Ανάπτυξης. Γιατί Πολλοί αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες προμηθεύουν με τα προϊόντα τους στις ευρωπαϊκές αγορές και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει και τους προμηθευτές από, ε, μη, ε, ε, από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι θέμα που μας αφορά, αφορά την Επιτροπή μας και έχω υποβάλει τροπολογίες. Αυτά ως εισαγωγή. Τώρα, ως ε, συντάκτης γνωμοδότησης, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό που η Επιτροπή ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και είναι καλό που συμπεριλαμβάνονται και οι μη Ευρωπαίοι αγρότες. Αυτό πρέπει να το καλωσορίζουμε και ορισμένες τροπολογίες που έχω υποβάλει κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Να ενισχύσουν το μήνυμα δηλαδή ότι αφορά η οδηγία αγρότες και παραγωγούς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που προμηθεύουν την Ευρωπαϊκή Αγορά. Εάν έχουμε διαφορετικά πρότυπα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πειρασμός στο σούπερ μάρκετ είναι να, θα είναι να προμηθεύονται από παραγωγούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να έχουμε ένα παιχνίδι επίσης όρης. Και νομίζω ότι η Επιτροπή Γεωργία στηρίζει την πρότασή μας αυτή. Οι άλλες τροπολογίες μου τώρα αποσκοπούν στην εναρμόνιση του κόστους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να υπάρχουν επίσης και καλοί ε, μηχανισμοί εφαρμογής των προβλεφθέντων στην νομοθεσία. Γιατί σίγουρα ε, η, η μάχη είναι άνηση οι παραγωγοί έχουν ένα μόνο αγοραστή, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και είναι πάρα πολύ δύσκολο να στραφούν εναντίον του και να υποβάλουν τα παράπονά τους και οι διεκδικήσεις τους. Επομένως, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους αγρότες ε, θα πρέπει να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση επίσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε παιχνίδι επίσης όρης και θα πρέπει εκ μέρους των αγροτών να μπορούν να ε, δρουν και συλλογικά όργανα και αυτά είναι τα βασικά μου μηνύματα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οκτώ τροπολογίες υποβάλλω μόνο και όλες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Και εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω, συντασσόμεθα απολύτως με τις προτάσεις και τις απόψεις της Επιτροπής για τα γεωργικά θέματα, της Επιτροπής Άγκρη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν τους σκιώδεις εισηγητές, έχουμε διάφορους ομιλητές. Ποιος θα ήθελα να μιλήσει για το θέμα αυτό η Μαρία Χόιμπουκ, καταγράφω τα αιτήματα, εσείς είστε αγρότης και είστε απολύτως ειδικοί να τοποθετηθείτε. Παρακαλώ. Ακριβώς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πράγματι με απασχολεί το θέμα, είμαι και σκιώδης εισηγήτρια στην Επιτροπή Γεωργίας, γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ακριβώς και εσύ Λίντα, επικρατώ και εγώ το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και επιδιώκει να τις ρυθμίσει όχι μόνο εντός αλλά και εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώντας τους ε, αγρότες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παράγουν προϊόντα για ε, κατανάλωση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πράγματι αθέμητος ανταγωνισμός, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν δίκαιες και σωστές τιμές για τους αγρότες. Θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό το ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες η παραγωγή πρέπει όντως στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία να έχουν την ε, δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματά τους. Και εμείς ως Επιτροπή Ανάπτυξης είμαστε αρμόδιοι και ε, οφείλουμε να φροντίσουμε ε, για την για τα δικαιώματα αυτά. Πρέπει να φροντίσουμε διάφορες ε, καταναλωτικές οργανώσεις, οργανώσεις παραγωγών ε, να ακούγονται, να δούμε πώς ε, μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τις, τους διάφορους συνεταιρισμούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, στην Μπουρκίνα Φάσο για παράδειγμα. Χρειάζεται επίσης ένα νέο σημείο επαφής το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε στην Επιτροπή αυτή. Τώρα, η Επιτροπή Γεωργίας έχει προτείνει ορισμένες βελτιώσεις με τις τροπολογίες της. Νομίζω πως αξίζει να στηρίξουμε τις τροπολογίες αυτές, οι οποίες αναφέρονται στους παραγωγούς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως δεν έχουν γίνει πολλά για τους παραγωγούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουμε να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους ε, αγρότες ε, στις χώρες εκτός ε, Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας, για αυτά τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διασφαλίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. κύριος Βέντα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εμείς στηρίζουμε τη γραμμή σας, την άποψή σας και σε αυτή την τροπολογία και στις υπόλοιπες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Και η κυρία Μέρκελ έχει πάει σε αυτές τις χώρες, τις Σενεγάλη μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αυτό είναι το θέμα, να δοθεί δημοσιότητα και να αναδειχθούν τα θέματα αυτά. Σε στηρίζουμε και σας ζητούμε να μεταφέρετε την προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα αντί για την Παρασκευή. Θα θέλαμε και εμείς να συντάξουμε κάποιες τροπολογίες και θα θέλαμε λίγο περισσότερο χρόνο. Επομένως, στηρίζουμε τις δικές σας και σας παρακαλούμε να μεταθέσετε την ε, καταληκτική προθεσμία για δύο-τρεις μέρες. Κοιτάξτε, ε, λέει η Πρόεδρος, η άκρη θα ψηφίσει την 1η Οκτωβρίου ε, και πλησιάζει ο καιρός. Επομένως πρέπει και εμείς να προλάβουμε να ψηφίσουμε. Είναι ήδη Τετάρτη. Τι, τι προθεσμία έχουμε την Παρασκευή, 12 το μεσημέρι ή 5 το απόγευμα. 6 το απόγευμα τη Παρασκευή να σα δώσω 6 το απόγευμα τη Παρασκευή, να σα δώσω 6 ώρε περισσότερε. σω το προσωπικό σα θα πρέπει να δουλέψει λίγο παραπάνω. Δεν μπορώ να αλλάξω, δεν μπορώ να δώσω το Σαββατοκύριακο και την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, θα το δεχτούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ο κύριο σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Από τη στιγμή που Έχουμε νέα αγορά και μάλιστα νέο νόμισμα. Συρώμαστε Μα έρνουν σε αυτή τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης όπου έχουμε μεγάλες ε, αγορές που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο ε, έχουμε προκηρύξεις και διαγωνισμούς σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή συγκέντρωση ε, σε ολίγους και δεν έχουμε ίδια νομοθετική ρύθμιση παντού. Άρα πρέπει κανείς να θέσει στον εαυτό του το εξής ερώτημα. Και εγώ ε, το γνωρίζω αυτό το θέμα γιατί έχω δουλέψει στην εγκατάσταση του Ιντερ Μαρσέ στην ε, Πολωνία, στην εγκατάσταση του Οσόν στη Ρωσία. Είναι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αυτές, γαλλικές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει κανείς να εξετάσει η ενιαία αγορά, η απαγκοσμιοποίηση, ο ανταγωνισμός, ο αγώνας για τη χαμηλότερη τιμή, όλα αυτά τα πράγματα που μας κατακλείζουν, ε, ε εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εθνών, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και δι των αγροτών. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυτή την παγκοσμιοποίηση και διαπιστώνουμε ότι ο μόνος τρόπος που έχουν για να επιζήσουν, να τα βγάλουν πέρα σε αυτό το σύστημα, είναι να μεταποιούν τα προϊόντα σε τοπικό επίπεδο και να τα πολλούν σε τοπικό επίπεδο. Μόνο έτσι μπορούν να τη βγάλουν. Και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο ε, της χαμηλότερης τιμής όπου ο παραγωγός πληρώνει, ακόμα και ο βιομηχανός. Πρόσφατα συμμετείχα σε ένα, στις συζητήσεις, δηλαδή πριν από τέσσερα χρόνια, με τους εκπροσώπους της γαλακτοβιομηχανίας για να επιβιώσουν. Μετά τους ήρθε το δίκαιο του ανταγωνισμού τα είχαν βρει. Ναι, ε, είχαν ένα, μια, ένα είδος συμφωνίας ε, για τις τιμές μεταξύ τους, αλλά ήταν για να μην το κλείσουν τα μαγαζιά τους τελικά. Και τελικά ήρθε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους έβαλε πρόστιμα και τους εξόντωσε. Δηλαδή, δεν είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων τις τιμές για να κερδοσκοπήσουν, αλλά για να απλά να επιβιώσουν. Πώς μπορούμε να έχουμε τοπική παραγωγή, τοπική μεταποίηση, τοπική πώληση. Αυτό είναι ο μόνος και ο καλύτερος τρόπος να επιτρέψουμε στους αγρότες να τα βγάλουν πέρα, να επιζήσουν και στους ντόπιου παραγωγούς. Ακόμα και τους μεγάλους και ακόμα και τις μεγάλες εθνικές βιομηχανίες τροφίμων. Μόνο έτσι μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Από εκεί και πέρα. Εγώ είμαι κατά του ελευθέρου εμπορίου πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε προνομιακές συμφωνίες με τους Αφρικανούς εταίρους και να έχουμε ε, σύντομους διάβλους. Δηλαδή χαίρομαι ότι πάω στο σούπερ μάρκετ και μπορεί ε, να αγοράσω μπανάνες ή καφέ ε, που προέρχονται από το δίκαιο εμπόριο, fair trade να πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή με τις προνομιακές σχέσεις και προνομιακές συμφωνίες που θα υπογράψουμε και που έχουμε υπογράψει. Δεν γίνεται να έχουμε έναν αγώνα για τη χαμηλότερη τιμή, για την συγκέντρωση ε, και για την καταστροφή των μικρών παραγωγών. Και πρέπει να ε, δώσουμε ε, το προνόμιο στην τοπική οικονομία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο τρίτων χωρών. Ναι, η Πρόεδρος, είναι απολύτως αληθές ότι γίνεται πολλής λόγος για την Αφρική, για τις θέσεις απασχόλησης στην Αφρική, για τους νέους Αφρικανούς που θέλουμε να μείνουν στη γη τους, να τη δουλέψουν, να προκόψουν, να έχουν δίκαια εισοδήματα για τα προϊόντα τους. Ο αγώνας για τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των ανταγωνιστικών μεγάλων αλυσίδων λιανικής στην Ευρώπη δεν βοηθά. Πράγματι πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα και δεν είναι το θέμα πάντοτε η χαμηλότερη τιμή. Εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ ε, πάνω στο ε, τομέα, ε, πάνω στη τιμή της μπανάνας και πρέπει να σας φέρω φωτογραφίες και διαγράμματα από τις αναλύσεις που έχουν γίνει για το τι απειροελάχιστα ψίχουλα παίρνει ο παραγωγός της μπανάνας από την τιμή στην οποία πωλείται. Τα σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει να ζητούν από τους αγρότες να πληρώνουν και για τα υπόλοιπα ε, και για τη συσκευασία. Δηλαδή Τώρα έχουν εξωτερικεύσει και έχουν αναθέσει όλα τα κόστη στου αγρότες και στους παραγωγούς οι μεγάλε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παλιά παρήγαγαν και τα έστελναν χήμα και ε, τα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ τα συσκεύαζαν και τα παρουσίαζαν στι προθήκε του. Τώρα θέλουν τη συσκευασία και όλα αυτά να τα κάνουν οι αγρότε και οι παραγωγοί και να, να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την τιμή του. Μένουν ψίχουλα. Δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο από ό,τι βλέπω. Η Επιτροπή είναι εδώ όμω. Κλούντιν Μέρκελ, δεν ξέρω να προφέρω σωστά το όνομά σα, ζητώ συγγνώμη, από τη Γενική Διεύθυνση για τα Γεωργικά Θέματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διορθώστε με παρακαλώ γιατί δεν πρόφερα σωστά το όνομά σα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για πρώτη φορά έρχομαι στην Επιτροπή σας. αμπληρωτής διευθυντής στην DG Agri και έχω αναλάβει αυτή την ε, πρόταση. Ευχαριστώ την Επιτροπή και σας που είστε οι συγκίτρια, Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη όπως τοποθετηθήκατε και στο σχέδιο γνωμοδότησης και η σύνταξη ε, αυτού του κειμένου ήταν κάτι το δύσκολο πήρε χρόνο και χαιρόμαστε που τελικά μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την προσπαθειά μας και να υποβάλουμε την πρόταση. Ε, είμαστε προσιλωμένοι στις αρχές που ενσωματώνει η υλοποίηση αυτή η πρόταση και θέλουμε να έχουμε στόχο το να υπάρξει πολιτική συμφωνία για το θέμα αυτό. Να κλείσει η συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους. Και πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας να έχει πάει αυτή η πρόταση στην επίσημη εφημερίδα. και θέλουμε βέβαια να μην ε, βάλουμε πάρα πολλές διατάξεις, πάρα, πολλές, πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτή την πρόταση γιατί τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα. Ε, όσο πιο πολλά είναι τα επίμαχα θέματα τόσο πιο δύσκολο είναι να υπάρξει συμφωνία και από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη και όλα αυτά να έχουν αίσια κατάληξη. Πρακτικό χαρακτήρα έχει αυτή η πρόταση, για την ε, ενημέρωση σε σχέση με τους προμηθευτές, σε σχέση με διάφορες χώρες, σε σχέση με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Πιστεύω ότι είναι εκείνη η στόχη που έχουμε εσείς και εμείς. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη γραφειοκρατία. και με την νομοθετική διαδικασία, με τον τριμερή διάλογο, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις στην οδηγία και να δούμε μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να οργανώσουμε αυτή την παροχή της πληροφόρησης και αυτό με τρόπο άτυπο. Να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να οργανώσουμε την δικτύωση ε, κρατών μελών Ευρωπαϊκής Επιτροπής των διαφορετικών υπηρεσιών τελικά να κάνουμε αυτό που κάνουμε και στον ε, ανταγωνισμό. Για την ε, στενή συνεργασία της Επιτροπής με τις αρχές ε, ανταγωνισμού των κρατών μελών. Κάτι άλλο τώρα το οποίο αναφέρεται στο σχέδιο κειμένου σας αφορά το ποιος δικαιούται να υποβάλει παράπονα καταγγελίες. Είπαμε για ενδιαφερόμενους φορείς, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η έννοια του ενδιαφερομένου. Να δούμε πως δεν θα πρέπει αυτό να αποτελεί μια ευκαιρία να δράσουν, να οργιάσουν οι κατ' επάγγελμα ενιστάμενοι και κατάγγελοντες. Κάποιος ανέφερε το ποιες είναι οι ευρύτερε συνέπειες της εμπλοκής των ε, γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αντισώμενες χώρες. Εμείς αυτό το οποίο προτείναμε θέλουμε να αποτελεί τμήμα της ε, ΚΑΠ. Θέλουμε να είναι κάτι που να βασίζεται στο άρθρο 43 της συνθήκης. Αυτό είναι ένα μόνο τμήμα μια ευρύτερης στρατηγική για το πώ θα δυναμώσει, πώ θα ισχυροποιηθεί η θέση η σε αυτή την υπόθεση των γεωργών να συνεργάζονται καλύτερα, να συνεργάζονται καλύτερα ε, είτε στα πλαίσια των συνεταιρισμών, των ενώσεων παραγωγών. Αυτούς θέλουμε να ενισχύσουμε. Προβλέπονται βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις από το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ε, έχουμε τον κανονισμό Omnibus, τώρα ισχύει. Ελπίζουμε ότι θα είναι πρακτική θετική εφαρμογή του Σακρατημέλη και επίσης τώρα υπάρχει η πρόταση να απαγορευτούν κάποιες αθέμητες πρακτικές, να έχουμε περισσότερη διαφάνεια στην τιμολογιακή πολιτική όσον αφορά διατροφική αλυσίδα. και ίσως με περισσότερη μελέτη επιπτώσεων μέχρι τα τέλη του έτους να έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα. Άρα δεν έχουμε εδώ μια παρέμβαση σημειακή, συγκεκριμένη. Πρόκειται για μέρος ευρύτερης προσέγγισης. Για να δούμε τώρα την νομοθετική διαδικασία, την τριμερή διάλογο με τα θεσμικά όργανα. Αυτό που θέλουμε να με χρονιά και να έχει γίνει η έγκριση κατά τη διάρκεια αυτή τη κοινοβουλευτική θητεία. Ελπίζουμε θα είσαι στο πλευρό μα σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήταν κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Και όσο τώρα να μην ξέρει κανένα τι συνέβη στην πρόταση αυτήν και να ξαναψάχνουμε να βρούμε το νήμα της χαμένης πρότασης μετά τις ε, εκλογές. Σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις Είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε στο Κοινοβούλιο, διότι είμαι ευρωβουλευτής πολλά χρόνια και θυμάμαι τις ε, γραπτές δηλώσεις, νομίζω τουλάχιστον πριν από δύο κοινοβουλευτικές θητείες, που ζητούσαν να αναλυφθεί δράση και τελικά δεν έγινε τίποτα ε, σε επίπεδο ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν η πίεση πρέπει να ε, συνεχίσει να ασκείται. Σε εθνικό επίπεδο να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει νομοθετική αντιμετώπιση, να υπάρχει μια προσπάθεια τέλο πάντων για εναρμόνιση. Και νομίζω πως τώρα υπάρχει η δυναμική για να γίνει επιτέλους κάτι. Τώρα, στο πλαίσιο των τριμερών διαλόγων, δεν ξέρω πώς θα συντονίσουν τα κρατημέλη τις διάφορες, διάφορους οργανισμούς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η Επιτροπή Γεωργίας είναι η αρμόδια επιτροπή και ε, σήμερα το πρωί συζητήσαμε και για ε, το fair trade και για το εμπόριο ανθών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει περιορισμός ή μιλάτε γενικά για γεωργικά προϊόντα. Κάθε συζήτηση τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εστιάσει στην λυσίδα τροφίμων. Διότι εκεί εντοπίστηκαν και τα προβλήματα. Επίσης, ε, έχουν συζητηθεί και άλλα γεωργικά προϊόντα, όχι μόνο στην ε, Κομάγκρη, όχι μόνο λοιπόν ε, λουλούδια, αλλά και υφάσματα, θα μπορούσε για παράδειγμα να συμπεριληφθεί και το βαμβάκι. Και νομίζω πως σημαντική θα είναι η ανάλυση μας για τις ε, σχέσεις ανάμεσα ε, στα διάφορα στάδια της παραγωγής. Θα ε, έχουμε ίσως νομικά προβλήματα για να συμπεριλάβουμε αυτά τα προϊόντα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Νομίζω πως εν ώψη εκλογών θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε αυτό. Είναι κάτι που μπορούν να καταλάβουν τόσο οι καταναλωτές όσο και ε, το ευρύτερο κοινό. Η προθεσμία ισχύει 31 Αυγούστου, Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα. Στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε την επόμενη φορά που θα συνεδριάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο σημείο 9. Συνάδελφοι, η κατάσταση εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Καταπιστευματικού Ταμείου Εκτάκτου Ανάγκης για την Αφρική. Όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ ήσυχα. Τώρα, συνάδελφοι, γνωρίζετε την ύπαρξη του καταπιστευματικού ταμείου. Δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Υπήρξε έκθεση ιδέα πρωτοβουλίας από τον Ιγνάτσιο Κοράο πριν από δύο χρόνια περίπου. Υπάρχει και ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό με πρόεδρο την Έλλη Σλάιν από τη δημιουργία του Καταπιστευματικού Ταμείου και έπειτα. Έχουμε προσπαθήσει, ασκώντας πίεση, να ε, ζητήσουμε και να λάβουμε μία θέση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Καταπιστευματικού Ταμείου. Η επόμενη συνεδρίαση του είναι στις 17 Σεπτεμβρίου. Επίσης, έγιναν και δύο αποστολές για να δούμε πώς χρησιμοποιείται το Ταμείο στην Αφρική. Η πρώτη αποστολή έλαβε χώρα στη Σενεγάλη το Φεβρουάριο που μας πέρασε και η δεύτερη στην Ουγγάντα το Μάιο. Εκεί είδαμε στην πράξη τη δράση του καταπιστευματικού ταμείου. Φυσικά η δράση δεν ε, ήταν και χωρίς διάφορα προβλήματα. Και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, να σας υπενθυμίσω ότι η πρόσφατη η πιο πρόσφατη μάλλον συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 500 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ε, παρακολουθούμε την χρήση του, του ποσού αυτού και σε γενικές γραμμές η αξία του καταπιστεύματος είναι 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλλον με συγχωρείτε, Αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Το σύνολο είναι 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 700 εκατομμύρια ευρώ για αναπτυξιακή βοήθεια και το συνολικό ύψος του καταπιστεύματος είναι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σκεπτικό πίσω από τη χρηματοδότηση ήταν πως η χρηματοδότηση θα ε, προέρχεται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα συμπληρώνουν ε, στο ε, καταπιστευματικό ταμείο. Η συνεισφορά μέχρι τώρα είναι 24,7 εκατομμύρια ευρώ, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Αλλά ο Μανουέλ ίσως έχει πιο ακριβείς πληροφορίες. Πολύ μικρό ποσοστό λοιπόν της χρηματοδότησης προέρχεται από τα κράτη-μέλη, κάτι που δεν είχε σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Θα δώσω όμως το λόγο στον Ιγνάσιο Κοράο, διότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες που πρέπει να συζητήσουμε και εκείνο ξέρει καλύτερα. Ήσουν παρόν Ιγνάσιο, σου δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο. Θα για να μας ενημερώσεις για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου ανάπτυξη. Θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, την Βερσέ από την ομάδα για την Αφρική, τον κύριο Κάι Κράιμπικ, αν προφέρω καλά το όνομά σας, για την ε, υπευθύνη για την Βόρεια Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα μας δώσει μια γενική εικόνα της κατάστασης και θα μας ενημερώσει για τις ε, πρόσφατες εισρωές κονδυλίων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ο λόγος της αύξησης του ταμείου αυτού θα μας πείτε... Θα μας πείτε εσείς μάλλον, αν γνωρίζετε από πού προέρχονται τα χρήματα, από ποιον προπολογισμό είναι κονδύλια τα οποία προέρχονται από κάποια άλλη γραμμή του προπολογισμού. Θα τα ακούσουμε όλα σε λίγο. Ο κύριος Βερσέ, λοιπόν, πρώτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της κατάστασης που έχει να κάνει με την εφαρμογή και υλοποίηση του καταπιστευματικού ταμείου. Έχουμε 3,9 δις ευρώ, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, που έχουμε, με τα οποία έχουμε περικοδοτήσει το ταμείο ως πόροι. Τα βλέπετε και στην οθόνη. Δεν ξέρω πώς να βγάλω αυτό το μικρό πλαίσιο που καλύπτει. Τέλος πάντων, 3,5 δις έρχονται από το προϋπολογισμό και από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και τα υπόλοιπα για να φτάσουμε στα 3,9 δις έρχονται από τα κράτη-μέλη. Έχουμε 71% από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, 17% από τον προϋπολογισμό της Επιτροπής, δηλαδή από το DCI και το ENI και 11% από τα κράτη-μέλη. Το DCI είναι το εργαλείο για την αναπτυξιακή συνεργασία και το ENI είναι το εργαλείο για την ευρωπαϊκή γειτονία. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθεια να συνεισφέρουν πιο σημαντικά και με πιο πολλά λεφτά στο καταπιστευματικό ταμείο. Με αυτά τα σχεδόν 4 δις ευρώ αποφασίσαμε να έχουμε 165 προγράμματα, 3,62 δις Δηλαδή 900 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν διαθέσιμα, δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί και προοριστεί για κάπου. 300 συμβάσεις ε, ε, έχουμε υπογράψει ύψους 1,6 δις, άρα το διακύβευμα παραμένει. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ώστε να πιο γρήγορα, αλλά να μην κάνουμε παρεκκλήσεις και να μην παρεκκλίνουμε από τους κανόνες που διασφαλίσουν την ποιότητα στις δράσεις μας. Ε, πρέπει να υπογράψουμε και να υλοποιήσουμε διάφορες συμβάσεις με τους διάφορους φορείς. Τρία είναι τα παράθυρα. Σε αυτά τα τρία δις 150 εκατομμύρια που αποφασίσαμε, βλέπετε εκεί την κατανομή του. Το μισό από, από το ποσό αυτό θα πάει για τη λίμνη του Τσάντ, το 1 τρίτο θα πάει στο κέρας της Αφρικής και τα υπόλοιπα στη Βόρειο Αφρική. Γιατί? Για τους εξής λόγους. Πρώτον, έχουμε με τις, τις κατανομές που έδωσε η αρμόδια Γενική Διεύθυνση για τη Βόρεια Αφρική. Και δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό ε, μέρος του αποθεματικού για, το, για τη λίμνη του Τσάντ, για την ε, επανένταξη και μαδενσωμάτωση μεταναστών που επιστρέφουν από τη Λιβύη και το να επιστρέψουν από τη Λιβύη και να ενσωματωθούν, αυτό στοιχίζει πολύ πιο ακριβά από, από ό,τι, ό,τι χρηματοδοτείται από το αποθεματικό για τη Βόρεια Αφρική. Αν μιλήσουμε για την κατάσταση στη Λιβύη, Έχουμε Αφρικανούς από τα μέρη κάτω από τη Σαχάρα, από τις χώρες του Σαχέλ και της Δυτικής Αφρικής και η επανενσωμάτωση και επανένταξή τους χρηματοδοτείται από το φάκελο για τη λίμνη του Τσάντα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ε, το γεγονός ότι θέλουμε να έχουμε πολύ καλή παρακολούθηση της χρήσης και αξιοποίησης των κονδυλίων, να έχουμε επιστροφή και ανατροφοδότηση, monitoring, αξιολόγηση και επανεκτίμηση το γρηγορότερο δυνατό. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει 41 παγκόσμιους δείκτες σήμερα και έχουμε και ένα εργαλείο για το reporting που λέγεται ICVO. Και έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα παρακολούθησης και μάθησης, monitoring και learning. Είναι το MLS, Monitoring and Learning System, σύστημα παρακολούθησης και μάθησης που θα εφαρμοστεί και στα τρία αυτά παραθυράκια στο κέρας της Αφρικής, στη Βόρεια Αφρική και στην λίμνη του Τσάντα. Έχουμε υπογράψει σύμβαση με την ίδια εταιρεία που θα τα κάνει όλα αυτά για να μπορούμε να έχουμε εκθέσεις που, εκθέσεις που θα συνδέονται με τα αποτελέσματα. Μπορεί κανείς ατέρμονα να μιλάει για το τι συμβάσει έχει υπογράψει και τι κονδύλια έχει δεσμεύσει, αλλά να μην έχει αυτά αποτελέσματα. Ενώ εμείς με τις συμβάσει αυτές θα μπορούμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα, θα μπορούμε να τα μετράμε και να τα αξιολογούμε άμεσα για να δούμε πώς ε, ε, διοχετεύονται τα λεφτά του καταπιστευματικού ε, ταμείου. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αξιοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες. 20.000 είναι οι δικαιούχοι 60% εκ των οποίων γυναίκες έχουν ε, ωφεληθεί από επαγγελματική κατάρτιση, για παράδειγμα. 46.000 μεταναστές και θύματα τράφικιν, παιδιά κτλ. έχουν δεχθεί βοήθεια στο πλαίσιο του φακέλου για το κέρας της Αφρικής. 2.000 άνθρωποι στις διοικήσεις στο κέρας της Αφρικής έχουν ωφεληθεί από καταρτήσεις ε, και εκπαιδεύσεις για το πώς θα διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές. Επομένως, δεν είχαμε τέτοιου είδους reporting για τις χώρες του Σαχέλ συνολικά. Αυτή τη στιγμή υπογράφουμε τις συμβάσεις, όμως έχουμε πολύ καλό reporting και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Θα σας δώσω κάποια νούμερα. 41.000 άνθρωποι στηρίχθηκαν στις χώρες του Σαχέλ, στις χώρες δηλαδή της Δυτικής Αφρικής, για να επιστρέψουν από τη Λιβύη ή που έχουν βρεθεί πάνω στους δρόμους των μεταναστευτικών ροών και ε, επέστρεψαν στις χώρες τους και έτυχαν στήριξης. 3.200 άνθρωποι έτυχαν ψυχολογική στήριξη, 4.300 άνθρωποι έτυχαν κοινωνική στήριξη σημαντικής, 5.740 ε, άνθρωποι έτυχαν οικονομικής στήριξης. Άρα έχουμε ε, νούμερα και στοιχεία ε, σε σχέση με την εταιρική σχέση που έχουμε με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Για εμάς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα είναι εκεί, απτά έρχονται και έχουμε αυτό το ε, σύστημα που μας βοηθά να τα αξιολογούμε και να τα παρατηρούμε. Έχουμε αξιοποίηση 41 δικτών, monitoring, σύστημα learning, μάθηση, δηλαδή να μαθαίνουμε για να αμέσως να διορθώνουμε και βλέπουμε αυτά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα. Έχουμε και τις κλασικές προσεγγίσεις για το monitoring και την αξιολόγηση που υιοθετεί πάντοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι συνδέεται με την αξιολόγηση και την ενδιάμεση αξιολόγηση αυτό το προγραμματίσαμε και το προγραμματίζουμε και για το 2018 και θα έχουμε τα αποτελέσματα για το 2019 γιατί η ενδιάμεση αξιολόγηση κρατάει πολύ. Αλλά έχουμε και το κλασικό ROM, Results Oriented Monitoring, παρακολούθηση που είναι προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα. Ξέρετε ότι Έχουμε και έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο για τις επιδόσεις μας που διενεργείται αυτή τη στιγμή και θα δώσει αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς. Τελευταία διαφάνεια για να δούμε την γενικότερη εικόνα, μια συνολικότερη εικόνα των προκαταρκτικών και προσωρινών αποτελεσμάτων, τα οποία μας φέρνει και μας δίνει το σύστημα ΑΚΒΟ και τα έχουμε επίσης και χάρη στην πρώτη έκθεση που έχει συνταχθεί και για τους τρεις τομείς, για τα τρία πεδία ή τους τρεις φακέλους αν θέλετε, λίμνη του Τσάντ, κέρας Αφρικής, Βόρειος Αφρική, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με τη μετανάστευση, αλλά καταπολεμούμε και τα εγκληματικά ε, δίκτυα και οργανώσεις. Για παράδειγμα, στο Νίγηρα έχουμε εξουδετερώσει και ε, ε, αδρανοποιήσει εγκληματικές οργανώσεις και έχουμε σώσει ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση με το μέσο της ερήμου όταν τους εγκαταλείπουν πάνω στη μεταναστευτική οδό. Ε, βλέπετε ε, πώς, πώς 44.000 άνθρωποι που ήταν σε ε, ευάλωτη κατάσταση έχουν βοηθηθεί κατά την άφηξή τους. Το 2018 και το 2019 θα είναι έτη στα οποία θα αφιερώσουμε τις προσπάθειές μας να έχουμε όσο να το περισσότερες πληροφορίες, απτές πληροφορίες για τα απτά αποτελέσματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Κλάιμπικ από την ε, Γενική Διεύθυνση Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Τιδιέ, σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ε, πω μια σύντομη εικόνα τι γίνεται για την Αφρική όσον αφορά το καταπίστευμα να αρχίσουμε με κάποια στοιχεία. Διαπιστώσατε ότι Έχουν 554 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα δεσμεύσει και 400 περίπου εκατομμύρια και αρχάς Ιουλίου έγινε μια συνάντηση και είπαμε ότι έχουμε τρία προγράμματα με 90,5 εκατομμύρια τα οποία έχουν εγκριθεί. Το σύνολο είναι πάνω από 50% του δεσμευθέντος ποσού και έχουμε εκταμιεύσει ήδη 80 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά πρόκειται να υπάρξουν και άλλες εκταμιεύσεις ε, μεγαλύτερα από εσάς Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Επίσης, να σας πω ότι όπως διαπιστώσατε, έχουμε 11% που θα καλύψουν τα κράτη-μέλη για την Βόρεια Αφρική. Έχουμε μεγαλύτερα ποσά 248,3 είναι τα εκατομμύρια που θα συμβάλλει ο γενικός προπολογισμός και 5,6 από τα κράτη-μέλη. Συνολικά άρχισετε μία ματιά το για 18 και το 19 έχουμε ένα κενό 75 εκατομμυρίων ευρώ και αποφασίσαμε να υπάρξει νέα συμβολή 148 εκατομμύρια ευρώ για την Βόρεια Αφρική. Πασμένο μήνα συμβούλες των κρατών μελών και άλλα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ θα είναι τα έργα τα οποία θα ακολουθήσουν για να καλυφθεί ένα τμήμα του κενού. σας παρουσίασε σχεδόν το σύνολο των αποτελεσμάτων που πετύχαμε για την Λιβύη έχουμε 44.000 μετανάστες και 55.000 προσώπων που χρειάζονται άμεση βοήθεια και περίπου 20.000 μετανάστες που έχουν τύχει αυτής άμεσης αρρωγής. UNCR, UNICEF, επίσης είναι η βασική μας ε, εταίρη και αν χρειαστείτε περισσότερα στοιχεία να σας τα παράσχω. Άρα, συνολικά, όσον αφορά την χρηματοδότηση από το EDF, θα να υπολογίσω, είναι περίπου 10%. 10% θα πάει στο καταπίστευμα. 71% όχι, όχι, ενώ από το σύνολο του προϋπολογισμού του EDF δεν είναι το 10%. γιατί αν δεν έχουμε περίοδο προγραμματισμού, αυτό θα πρέπει συνάδελφοι να λάβουμε υπόψη, γιατί είναι πολλά τα χρήματα ο πλευρά CDF που θα πάνε σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν κάτι πια πάρα πολύ σημαντικά έργα στην Ουγγάντα και πρόκειται για πολλά χρήματα που προέρχονται από αυτά τα ταμεία και πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Έχουμε τον Ιγνάτσιο Κοράο, που είναι ο εισηγητής μας. Συμμετάσχει και στο στρατηγικό συμβούλιο. Να δούμε πώς θα υπάρξει η ενημέρωσή μας για τις συναντήσεις της 17-18 ε, Σεπτεμβρίου. Πέφτει Παρασκευή, οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Τι λες, Σε ευχαριστώ, Λίντα. Και Ευχαριστούμε για την Επιτροπή, για την εισήγηση, για τις εξηγήσει συμμετέσχων στο Συμβούλιο και ζητήθηκε αυτό σε εκείνη την έκθεση που είχα αναλάβει ήταν σημαντική αυτή η εμπειρία γιατί έτσι είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω εκ του πως λειτουργεί αυτό το καταπίστευμα παρακολούθηση και τη συζήτηση για την κατανομή των ε, πόρων. Και υπήρξε βέβαια κάποιος δισταγμός από πλευράς κρατών μελών όσον αφορά την συνεισφορά τους ή στο καταπίστευμα και πρώτα-πρώτα νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να δίνουν προτεραιότητα σε ό,τι έχει σχέση με δικά τους τοπικά, γεωγραφικά, ούτως υπήν συμφέροντα. Και το πρόκειται τώρα για ένα καταπίστευμα, ένα ταμείο που πάνε πάρα πολλά χρήματα. Αυτά τα οποία μας ε, παρουσίασε η Επιτροπή και έχουμε για τα συστήματα της ε, εποπτείας δεδομένα. Και έχουμε επίσης και τη σύσταση 15 του 18 του ελεγκτικού συνεδρίου για το πώς θα είναι αποτελεσματική η κατανομή των ε, πόρων. Ε, αυτά θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη για τη συνεισφορά τους. Πέντε από τις έξι προτεραιότητες συζητήθηκαν εκεί στο Συμβούλιο όσον αφορά το τι θα γίνει με την ε, μετανάστευση, πώς θα αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίε και κάτι άλλο που εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι αυτά τα έργα, αυτά τα προγράμματα ε, σε υπηρεσίες βάσης και αυτό έχει να κάνει και με τις αιτίες της μετανάστευσης, γιατί εάν ε, διαθέτουμε τρόφιμα, εάν δίνουμε τη βασική αρρωγή σε ε, κάποιους πληθυσμούς που είναι στριμωγμένοι, ε, αυτό είναι βοήθεια. Αυτό δεν είναι παρέμβαση στις αιτίες της μετανάστευσης. Επομένως, εάν μετακινούμε από το Ταμείο Ανάπτυξης κάποιους πόρους, θα πρέπει να δούμε το πώς θα δημιουργηθούν όροι, υπόθεσεις οι όροι και προϋποθέσεις τέλος πάντων για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Πέραν του να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τη μετακίνηση εκατομμυρίων από τη μία ήπειρο στην άλλη είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και αυτό θα πρέπει να δούμε για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και επίση είναι θέμα διεθνούς συνεργασίας, δεν είναι θέμα μόνο της Επιτροπής μας και θα πρέπει να δούμε το ότι πρόκειται επίσης για θέμα υψή τη προτεραιότητα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποπτεία, απόσπαση αποτέλεσμάτων, ανάπτυξη συγκεκριμένη, συνθήκες διαβίωσης. Εκεί στις χώρες που γίνεται κυρίως η διαμετακόμιση, η διέλευση όλων αυτών των ε, ανθρώπων που θα καθορίσει και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να είμαστε επομένω πολύ συγκεκριμένοι στο τι θα κάνουμε, ποιους δείκτες ανάπτυξης θα μετέλθουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε. Τέλος πάντων, ε, έχουμε τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο είναι η μετανάστευση. Και θα πρέπει και αυτά να τα σπαστούν τα μέλη. Πάντως τελικά δεν ε, υπήρξε συμφωνία όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά. Άρα τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμα δεν διατέθηκαν οι αναγκαίοι πόροι. Είναι θέμα του κοινωτικού προϋπολογισμού. Έλλη, ασχολείσαι με τη μετανάστευση. Θες κάτι να μας πεις, έχεις κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το καταπιστευματικό ταμείο εκτακτή ανάγκη για την Αφρική δημιουργήθηκε πριν από περίπου τρία χρόνια και από τότε η Επιτροπή μα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των διαφορών μέσων και την ε, κατανομή των σχετικών κονδυλίων. Τον Φεβρουάριο δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασία τη Επιτροπή Ανάπτυξη έτσι ώστε να δώσει ένα πλαίσιο στην παρακολούθηση και τον έλεγχο ε, στον ε, τομέα της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας για τη μετανάστευση. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητε του Καταπιστευματικού Ταμείου για την Αφρική, που αποτέλεσε και αντικείμενο του ελέγχου μας πέρυσι, στόχος μας ήταν να επαληθεύσουμε ότι τα δύο αυτά ταμεία δεν χρησιμοποιούνται αντίθετα από τους στόχους τους. Δημιουργήθηκαν λοιπόν ανησυχίες για την πιθανή ανακατεύθυνση κονδυλίων που προορίζονται για την ανάπτυξη σε διαχείριση συνόρων, σε μετανάστευση και αυτό υπονομεύει τους ε, στόχους της ε, ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το ταμείο αυτό είναι ένα μέσο το οποίο υποτίθεται πως στόχο έχει να συνδράμει στην καταπολέμηση των αιτίων μετανάστευσης. Και η κύρια έμφαση που δίνει είναι, είναι στην επιστροφή των ε, ανθρώπων που έχουν φύγει από τις ε, χώρες τους, από τις πατρίδες τους, ε, λόγω φτώχειας, λόγω πείνας, ε, πολέμου κτλ. Επίσης υπάρχει υπάρχει διαβούλευση με τοπικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Το καταπιστευματικό ταμείο ναι μεν εγγυείται δια... Ε, αυτή την συνεργασία, όμως εις βάρος της διαφάνειας και της ε, λογοδοσίας. Το Κοινοβούλιο έχει περιορισμένο έλεγχο. Έχει μεν κληθεί να συμμετέχει στη συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτό είναι θετικό, όμως ήταν πολύ δύσκολο ε, να παραστεί Εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα λόγω συναντήσεων σε εβδομάδα ολομέλεια ή πράσινη εβδομάδα κτλ. Οι διάφορες επιτροπές αποφασίζουν για το ποια project θα χρηματοδοτηθούν και αυτό είναι και το σημαντικότερο. Πρέπει να καταλάβουμε με ποια κριτήρια επιλέγονται τα διάφορα ε, έργα προς χρηματοδότηση. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι η πλειοψηφία των ε, χρηματοδοτούμενων έργων υλοποιούνται από κρατικούς ε, φορείς. Υπάρχει γενικότερα ένας δισταγμός των κρατών μελών να συνεισφέρουν κονδύλια στο καταπιστευματικό ταμείο. Ορισμένα κρατημέλη αναφέρονται σε αρνητικές ε, επιπτώσεις. Στην περίπτωση του Νίγηρα, για παράδειγμα, πως ε, αποδομούμε τον ε, εμπορικό ιστό χωρίς να παρέχουμε κάποια εναλλακτική λύση και αυτό αναπόφευκτα θα έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της χώρας και στην ε, νομιμότητα των αρχών της περιοχής. Επίσης, θέλετε πως υπονομεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, ανθρώπων στην περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι η οικονομία χωρών της Αφρικής στηρίζεται και βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία και είναι πολύ σημαντικό να μην υπονομευτεί αυτό. Έπειτα, Λιβύη. Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία στοχεύουν στην ε, στήριξη των ε, αρχών, για παράδειγμα τα έργα που ε, στηρίζουν το έργο της ακτοφυλακής υπονομεύουν πολλές φορές το διεθνές δίκαιο. Σημειώνεται παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την ακτοφυλακή της Λιβύης. Υπάρχουν λοιπόν αρνητικές επιπτώσεις που θα επιδεινώσουν την ήδη θραυστή κατάσταση στην Λιβύη. Μετά, σε άλλες χώρες, στην Ουγκάντα. Υπάρχουν διάφορα έργα στήριξης της επαγγελματικής κατάρτισης με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Μας προειδοποιούν αρκετές χώρες πως ε, δεν χρησιμοποιούνται τα χρήματα έτσι όπως πρέπει. Ε, για παράδειγμα, υπάρχουν αναφορές σε έκτακτες ανάγκες χωρίς να ε, δίνονται λεπτομέρειες σε γενικές γραμμές αυτό που πρέπει να... Σε αυτό πρέπει να δώσουμε βάση είναι στους μακροπρόθεσμους ε, στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εξωτερικεύσει την ε, φύλαξη των συνόρων της και αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν κονδύλια που χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια ευρώ που έχουν διατεθεί για αυτό το σκοπό από άλλα ταμεία και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να μην εγκαταλείπουμε τη, την προσπάθεια προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, προς όφελος εσωτερικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν με αυτόν τον τρόπο θα συνεισφέρουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και θα ε, δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους Αφρικανούς. Δεν είμαι τόσο σίγουρη ε, και από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα νομίζω πως η κατάσταση είναι ανησυχητική. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει πολλοί συνάδελφοι το λόγο. Πέντε. Ο κύριος Τσέλερ, η κυρία Σαρτζεντίνη, ο κύριος Σάφαουζερ, η Τέστα Χιμένεθ και η Σεσίλ Κέγγε. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Όχι. Κύριος Τσέλερ, λοιπόν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πολύ σωστά συζητάμε αυτό το θέμα σήμερα και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που συνεργάζονται για αυτό το θέμα. Το καταπιστευματικό ταμείο στόχο έχει γρήγορη παροχή βοήθειας ε, για ε, θέματα ανθρωπιστικής ε, βοήθειας και για την καταπολέμηση των αιτίων διαφυγής από τις χώρες προέλευσης. Το καταπιστευματικό ταμείο λοιπόν δημιουργήθηκε με πρόσθετα κονδύλια και υπάρχει ε, διοχέτευση κονδυλίων από άλλα ταμεία. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό. Ε, το, ένα, το μεγαλύτερο ποσοστό του καταπιστευματικού αυτού ταμείου προέρχεται από ε, χρηματοδότηση από άλλα ταμεία, από το Ειδικό Ταμείο Ανάπτυξης, ε, νομίζω το μεγαλύτερο μέρος είναι από αυτό, 11% από τα κρατη όπως ακούσαμε. Επίσης, τα κράτη-μέλη όταν δίνουν χρήματα ζητούν και αποτελέσματα και έλεγχο αυτών. Τώρα, το καταπιστευματικό αυτό ταμείο διοικείται όχι άμεσα από εμάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μάθω τι συμβαίνει με τη διοίκηση, ε, πόσο κοστίζει η διοίκηση του καταπιστευματικού ταμείου. Και επίσης, το σύνολο ε, της χρηματοδότησης, το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης που προέρχεται από το Ταμείο Ανάπτυξης. Τι μακροπρόθεσμους στόχους έχει. Υπάρχει προγραμματισμός μακροπρόθεσμος, περιφερειακός, ε, τοπικός, εθνικός ε, και ποια η σύνδεσή του με, το, με τα διάφορα έργα που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί μέλος, ε, μέρος της Συμφωνίας του Κοτονού ε, για συνεργασία με τα κράτη εκείνα που, έχουν, που την έχουν υπογράψει και έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες συνεργασίας και ανάπτυξης. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται σε χώρες και σε περιοχές όμως ε, οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού. Γι' αυτό λοιπόν ε, οι ερωτήσεις μου, πόσο μας κοστίζει το όλο εγχείρημα. Ποια είναι τα ποσοστά απορρόφησης. Μας λέτε πως είναι χαμηλά. Εγώ έχω διαβάσει και μία έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία ε, τα ποσοστά απορρόφησης ε, έχουν να κάνουν περισσότερο με διοικητικό κόστος. Και τα ποσοστά απορρόφησης επίσης ε, είναι μικρά και η απορρόφηση γίνεται πολύ αργά. Το θέμα σε ένα, και το ζητούμενο σε ένα καταπιστευματικό ταμείο είναι όλα αυτά να γίνονται γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. εξοδεύουμε το 10% του EDF στο καταπιστευματικό ταμείο, το 10% του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Πόσα όμως από αυτά τα χρήματα προορίζονται για την αντιμετώπιση των ε, βασικών αιτιών για τη μετανάστευση και ποιο μέρος από αυτά τα χρήματα δίδεται για την προστασία των συνόρων και τη μικροδιαχείριση σε επίπεδο καθημερινό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δούμε αυτά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν και πολλά που να είναι υπέρ του αναπτυξιακού σκέλους. Μιλούν, ε, χρησιμοποιούν τα κονδύλια όλο και περισσότερο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών την καθημερινή. Ενώ εγώ νόμιζα ότι κάναμε και αναπτυξιακή συνεργασία με τέτοια χρήματα. Μετά την επιστροφή σας από την Ουγκάντα, Λίντα, και μετά τον έπαινο των προγραμμάτων που είδατε εκεί να εφαρμόζονται, τίθεται το ερώτημα τι γίνεται με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των project αυτών δεν μπορεί κανείς να τρέχει αναπτυξιακά προγράμματα με πολύ βραχία χρηματοδότηση που θα λήξει γρήγορα. Εάν λοιπόν παρατηρείτε ότι υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης και είναι μακρά η συζήτηση που μας περιμένει και για το μέλλον της χρηματοδότησης, τότε μπορείτε να απαντήσετε ίσως στο εξή ερώτημα. Πώς θα διασφαλίσετε, πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα project που στοχεύουν προς την ανάπτυξη και προς την εξάλληψη των πρωταρχικών αιτιών της μετανάστευσης θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται και με την έλλειψη χρήματος πώς θα λειτουργήσετε και ποια είναι η διαφοροποίηση που κάνετε μεταξύ Τη εξάλληψη των βασικών αιτιών της μετανάστευση και της καθημερινής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες ιδέες για το ε, ποιο μέρος της χρηματοδότηση πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικές κυβερνήσει και σε ποιο μέρος πηγαίνει στις μη κυβερνητικέ οργανώσει, είτε ντόπιε είτε διεθνεί. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα ερωτήματα. Θα επανέλθουμε. Ο κύριος Σαφχάουζα, παρακαλώ. Ναι, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για το καταπιστευματικό ταμείο. Ήμουν υπέρμαχος αυτού του ταμείου και τώρα έχω αρχίσει να αναθεωρώ. Γιατί είδα πόσο λίγο αποτελεσματικό είναι στην, για παράδειγμα στην κεντροαφρικανική δημοκρατία σε μια χώρα. Νομίζω ότι καλούμαστε να κάνουμε μια επιλογή. Είτε δίνουμε επίγουσα βοήθεια και πρέπει να το κάνουμε, για την επίγουσα η κατάσταση και άρα στηριζόμαστε στις μη κυβερνητικού οργανισμούς, είτε είμαστε στο σκέλος ασφάλεια και ανάπτυξη, άρα πρέπει να στηριχθούμε στις κρατικές δομές. Και δεν μπορεί τίποτα να γίνει χωρίς να υπάρχει κράτος. Και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι κράτος νόμιμο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με νόμιμες θεμητές απολύτως λογικές εκλογές. Άρα, για την χώρα αυτή μιλώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολύ συγκεκριμένη περίπτωση αυτή της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας. Σε θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης δεν σταθήκαμε ικανοί να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ασφάλειας που είναι ε, απολύτως απαραίτητες. Η κατάσταση ασφαλείας έχει υπονομευτεί, έχει υποβαθμιστεί, έχει χειροτερεύσει. Η Ρωσία τελικά παρέμβει παρενέβηκε και με τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών και να μην ξεχνάμε να το λέμε αυτό και ε, τρόποντινά νομίζω ότι φαινόμαστε γελοί. Και αντιθέτως με αυτά που λέει η συνάδελφος, εγώ πιστεύω ότι είναι απολύτως αδύνατο να λυθούν τα προβλήματα ασφάλειας και ανάπτυξης εάν δεν στηριχθούμε στα κράτη. Αν αφήνουμε το κράτος να κάνει ό,τι θέλει, θα εξατμιστούν τα κονδύλια. Εάν στηρίζουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν ε, δίνουμε βοήθεια για ανάπτυξη, αλλά δίνουμε βοήθεια για επίγουσες περιπτώσεις. τώρα, πρέπει να έχουμε παράλληλες δομές με διαδικασίες, παράλληλες με τις κρατικές διαδικασίες και να απελευθερώνονται τα κονδύλια αναλόγως με την πρόοδο και με τη συμφωνία των τοπικών εκπροσώπων μας οι οποίοι δεσμεύονται καθ' τη διάρκεια της διαδικασίας και δεσμεύονται και για την αίσια έκβαση του προγράμματος. Εγώ όταν διαχειριζόμουν project πήγαινα ο ίδιος επί τόπου και έχω τη μύτη μου παντού μέχρι εσώτου να βεβαιωθώ ότι τα πράγματα γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Και βλέπω ότι δεν είναι αυτή η περίπτωση εδώ, δεν κάνουν το ίδιο. Οι ντόπιοι εκπρόσωποι ε, παίζουν το δικό τους βιολί και συνεννοούνται με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτά για την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Τώρα για τη λίμνη του Τσάντα. Στην ίδια κατάσταση, στο Μάλι. Το Μάλι, επίσης στην ίδια κατάσταση στο Μάλι. Έχει υποβαθμιστεί, έχει χειροτερεύσει, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Ό, τα αποτελέσματά μας είναι η γελία. Επομένως, κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και θα πρέπει να συντάξουμε ένα πρόγραμμα μαζί με το εκάστοτε κράτος, εάν αυτό είναι απαραίτητο, να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή του και δεν πρόκειται για νέο απικιοκρατία ή κάτι τέτοιο, είναι για μια ουσιαστική εταιρική σχέση. Και ε, χωρίς αυτό δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα και οι δείκτες σας δεν σημαίνουν τίποτα και δεν είμαστε στο ύψος των περιπταστάσεων. Άμα δείτε ε, την αποσταθεροποίηση και τα μεγέθη, τα δικά σας νούμερα είναι γελία. Ε, και Περνάτε το χρόνο σας να παίζετε με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και δεν ασχολείστε με το σκέλος της ασφάλειας και της ανάπτυξης που είναι απολύτως απαραίτητη για τις χώρες αυτές. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο. Μείναμε με την επισημία, αλλά το στομάχι αδιανό. Ε, δεν θα πρέπει να μείνουμε κολλημένοι στις τρευλώσεις του παρελθόντος. Η αποτελεσματικότητα δεν ε, είναι παρούσα, απουσιάζει. Δεν σας κρύβω την απογοήτευσή μου. Εγώ ήθελα να εμπλακώ προσωπικά στο θέμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, αλλά αποφάσισα να απέχω γιατί η ανασφάλεια έχει ενταθεί, έχει οξυνθεί. Ο πρόεδρος της χώρας αυτής στράφηκε προς τη Ρωσία τελικά και θα προτιμούσα εμείς να είχαμε καλύψει αυτό το χώρο. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον της Ρωσίας, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Ρωσία, αλλά εμείς χάσαμε την ευκαιρία και αυτό στράφηκε προς τη Ρωσία στη συνέχεια και είναι μια πραγματικά πολύ χαμένη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Μήπω οι συνάδελφοι μπορούν να μιλήσουν για το Ταμείο του Μπακού, Μπέκου Φαντ. Είναι κάποιο εδώ. Ο πρέσβης θα έρθει να μας δει την επόμενη εβδομάδα εάν θέλετε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό. Εν πάση περιπτώσει προχωρούμε στην Τερέζα Χιμένεθ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε και να τονίσω κάποια πράγματα τα οποία κάπως με ανασυχούν. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ταμείο αυτό. Απαραίτητο και δεν μας δίνει τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Δεν φέρνει τους καρπούς που θα έπρεπε να έχει φέρει. Νομίζω ότι από εδώ, από πλευράς Ευρώπης, κάναμε μια πολύ κακή πολιτική επικοινωνία. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής, ο μεγαλύτερος συνεισφέρον στο κόσμο, στην αναπτυξιακή βοήθεια και όταν μιλούμε για τη μετανόστευση όλοι λένε δεν κάνει τίποτα η Ευρώπη, το πρόβλημα είναι από την Ευρώπη πρέπει, πρέπει να δουλέψει στις χώρες προέλευσης και δεν το κάνει και η πολιτική στις, ε, στα εθνικά κανάλια και σε εθνικό επίπεδο συνεχώς λένε ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα στις χώρες προέλευσης και δεν έχουν ιδέα ούτε για, αυτή την, ε, για αυτό το ταμείο, ούτε για την ύπαρξή του, ούτε για την ύπαρξη όλων των δράσεων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, ασκήσουμε καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική, να διαδώσουμε περισσότερο τα νέα μας και τα αποτελέσματά μας και τις δράσεις μας, γιατί η κοινή γνώμη δεν έχει ιδέα για το πόσο παρόντες είμαστε και πόσα χρήματα δίνουμε στην Αφρική. Πράγματι, μεγάλο μέρος των χρημάτων πηγαίνει ε, στις δράσεις ασφάλειας, αλλά είναι και αυτό απαραίτητο. Πρόκειται για failed states, για αποτυχημένα κράτη. Και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, για παράδειγμα, ούτε εμεί δεν μπορούμε να πάμε. Και οι δικοί μας πρέπει να δράσουν για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από τη Σομαλία και αντίστροφα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που τρέχει ένα project ε, και ε, έρχεται ένας δικτάτορας οποιοδήποτε τα καταστρέφει όλα και ο αγρότης που είχε βοηθηθεί και είχε αρχίσει να ροντάρει τέλο πάντων την αγροτική του δραστηριότητα πρέπει ξαφνικά να τα αφήσει όλα και να φύγει, να πάει στη διπλανή χώρα να γλιτώσει. Δεν είναι μόνο το οικονομικό το θέμα και δεν είναι και αλήθεια αυτό στην Ιγυρία και στην Κάμπια δώσαμε πολλά χρήματα για την εκπαίδευση και την ε, ε, απασχόληση των νέων. Δώσαμε πάρα πολλά χρήματα για την καταπολέμηση της ε, εμπορίας ανθρωπίνων όντων, για το τράφικιν. Και στη δική μου περιφέρεια, στην Ανταλουσία. Είμαστε οι Ανταλουσιάνοι στην παραλία και βλέπουμε να έρχεται στο Τσικλάν, στον Μπαρμπάτε, παντού, να μπαίνει ε, η βάρκα το ε, δουλεμπορικό και να ε, ξεφορτώνει τους ανθρώπους και μάλιστα να μπαίνει με τεράστια ταχύτητα με κίνδυνο και για τους λουόμενους. Να έχουμε βεβαίως περισσότερους πόρους και να τους διαφοροποιήσουμε γιατί υπάρχουν επίγουσες καταστάσεις, υπάρχουν επίγοντα περιστατικά, υπάρχουν έκτακτα περιστατικά και δεν μπορούν όλα να τα βάλουμε στο καλάθι ενός μόνο ταμείου. Πρέπει να επινοήσουμε δράσεις και σε πιο, με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι χώρες αυτές έχουν φτώχεια ε, δεκαετιών και παραπάνω. Δεν μπορούμε να τη λύσουμε αυτή ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Να μελετήσουμε καλά πώς θα λειτουργήσουμε, πώς θα ε, ε, λύσουμε τα επίγοντα θέματα και να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα ε, να φανεί περισσότερο αυτό που κάνουμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πράγματα. Γιατί είναι άδικο να νομίζουν ότι δεν κάνουμε τίποτα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Τερέζα. Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, αλλά έχετε δίκιο. Υποτίθεται ότι ήταν Ταμείο αντιμετώπιση Επιγόντων Θεμάτων και απλά μένει μόνιμο και μόνιμο είτε. Η Φεντερίκα Μογκερίνη το έχει πει ότι είναι ένα μόνιμο φαινόμενο και θα πρέπει να έχουμε μόνιμα προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας πει. Ποιο κομμάτι πάει στο αναπτυξιακό σκέλος και ποιο μέρος των χρημάτων πάει στο σκέλος της ασφάλειας και της διαχείρισης των επιγόντων παριστατικών σε καθημερινή βάση. Ο κύριος Γκένγκια. Ο Σεσίλ. Ή Σεσίλ Γκένγκια ξέρει πολλά. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ Λίντα. Θέλεις να λάβω το λόγο για αυτό το καταπίστευμα. Και Τελικά είναι έτσι είναι. Πρόκειται για ταμείο καταπίστευμα επίγουσας φύσης, επίγουσες καταστάσεις. Ε, και βέβαια είναι το θέμα των ε, ε, αιτιών της μετανάστευσης, το θέμα του τι θα κάνουμε την ανάπτυξη και τι θα πρέπει, αν δεν τα καταλάβουμε καλά αυτά τα πράγματα, να πέσουμε σε κάποια παγίδα στο ότι αυτό το καταπίστευμα μπλοκάρει κάποιους που θέλουν να φύγουν από τη χώρα ε, προέλευσης και δεν μπορούν να πάνε στις ε, χώρες διαμετακόμισης για να φτάσουν στην ε, Ευρώπη. Βέβαια, εγώ δεν θέλω τέτοια προσέγγιση, πρέπει να σας το πω. Όμως, με αυτό το ταμείο προχωρήσαμε σύμφωνα με κάποιο σκεπτικό, γιατί βλέπουμε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα δύσκολο να έχουμε ενιαία άποψη για όλες τις χώρες που καλύπτει ε, αυτό το ταμείο. Μαλή, Σενεγάλη, Μπουρκίνα Φάσο, Σαχέλ. Υπάρχουν θετικά, αλλά υπάρχουν και αρνητικά από αυτή την ε, κατάσταση. Και με αφετηρία την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν φτάνει αυτή η πρικοδότηση δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις έτσι, ε, έτσι μια αλλαγή. Χρειάζεται μια αυθεντική πολιτική που να βοηθάει ε, για έργα, προγράμματα ανάπτυξης ε, για τα κρατή-μέλη να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά. Τώρα όσον αφορά τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες επιτόπου, το καταπίστευμα κατά τη γνώμη μου δεν έχει τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των διαχειριζομένων και από την άλλη μεριά των τοπικών αρχών. Έτσι θα πρέπει να δούμε πώς από το μηδέν θα έχουμε έργα και προγράμματα ε, και πώς δεν θα έχουμε επικαλύψεις με ήδη φυστάμενα προγράμματα και έργα. Επίσης δεν υπάρχει συντονισμός ε, σε σχέση με άλλα αναπτυξιακά προγράμματα. Άρα σε αυτό θα πρέπει να πασχίσουμε, να δούμε πώς θα υπάρχει περισσότερη ανθεκτικότητα του καταπιστεύματος, πώς θα χρησιμοποιηθεί ως καταλήτης. Δηλαδή να δούμε το πώς θα έχουμε συνέργεια μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων, να τα ενισχύσουμε και επομένως να δούμε το πώς θα υλοποιηθούν οι προσπάθειες αυτού του καταπιστεύματος επιτόπου. Και Όταν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις όπως στη Λιβύη, δύσκολο να μιλούμε για κατηγορίες ε, ε, δικαιούχων. Ε, πολλές φορές αυτοί που θέλουν να εμπλακούν αλλάζουν ιδιότητα από το βράδυ μέχρι το πρωί. Και τα προγράμματα εκτός του κατά πιστεύματο θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια σε σχέση με το περιβάλλον και σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους και την διαφάνεια. Προστασία του περιβάλλοντος. Εκεί θα πρέπει να κατατείνουν. Να το προσέξουμε αυτό. Όχι στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στη ρήπανση. Πολλές φορές αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για κάποια προγράμματα. Οπότε έχει καλός αυτό το καταπιστεύμα αλλά θα πρέπει να το θωρακίσουμε για τους πόρους, για τον συντονισμό επιτόπου και να δούμε και πάλι ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο συγκροτήθηκε. Να μην θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιούμε το καταπίστευμα για να φρενάρουμε τον κόσμο ε, στη χώρα προέλευσης ή στη χώρα διμετακόμισης. Δεν θέλουμε τα όρατα τείχη να ενισχυθούν. Θέλουμε με αυτό το εργαλείο να κάνουμε κάτι για τις αιτίες της μετανάστευσης και ο κόσμος νυφάλια να μπορεί να διαλέξει αν θέλει τι θα κάνει φεύγοντας από τη χώρα τυχόν, από τη χώρα της προέλευσης. Ας λάβουμε υπόψη επομένω και αυτό το ηθικό στοιχείο. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και να τα προσέξουμε επιδέχεται βελτίωση η κατάσταση, αλλά μόνο μέσω της συνεργασίας μας. Yeah, thanks. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε ένα θέμα πριν την συμφωνία για το Κοτονού και ένα άλλο θέμα για το Ταμείο Συλλού και Μετανάστευσης. Αν θέλετε λοιπόν να απαντήσετε, παρακαλώ λίγο σύντομα. Δεν ξέρω ποιος από εσάς θέλει να αρχίσει. Ο κύριος Βεξέ, Επίσης, ε, συνάδελφοι, σχετικά με την συνεισφορά των ε, κρατών μελών. Να σας πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτές τις συναντήσεις, η Επίτροπος Μογκερίνη υπενθυμίζει τα κρατημέλη να συνεισφέρουν ε, και τα κράτη-μέλη θεωρούν πως ε, τα χρήματα αυτά που είναι στο καταπιστευματικό ταμείο, ε, στο Ταμείο Ανάπτυξη είναι δικά τους, άρα έχουν συνεισφέρει. Ίσως λοιπόν ε, θα πρέπει εσείς να ασκήσετε πίεση στους υπουργού σας των οικονομικών για να συνεισφέρουν περισσότερο. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε για τα μεγάλα κράτη-μέλη, γιατί έχουμε 25% αυτού του καταπιστεύματος τα οποία καλύπτονται. Ε, ούτως ώστε αυτοί που δεν μπορούν να βάλουν χρήματα να καλύπτονται. Επίσης ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά τους βουλευτέ για την ανάλυση, για την πλαισίωση του θέματος, για όλα αυτά τα οποία είπατε είναι σημαντικά, θα βελτιώσουμε την πρότασή μας και ε, όλα αυτά δείχνουν το πόση σημασία αποδίδεται στο θέμα. Επομένω, ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα του θέματος της ανάπτυξης, θεωρούμε ότι 100% του καταπιστεύματος ε, επιδέχεται και περνάει από οικονομικό έλεγχο. Το σύνολο, επομένως, των πόρων διατίθεται για την ανάπτυξη. Τώρα, όσον αφορά την ε, ασφάλεια όσον αφορά τα σύνορα και αυτό καλύπτεται. Έχουμε επομένω μια κλασική προσέγγιση αναπτυξιακή. 50% του ταμείου πάνε στην απασχόληση και στην θωράκιση και ισχυροποίηση των πιο ευάλωτων 30% για τη διαχείριση της μετάσταση και 20% για την πρόληψη των συγκρούσεων και την ασφάλεια. Κλασική προσέγγιση έχουμε όταν είναι 50-50 η διάθεση των πόρων και επομένως ε, συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι στόχοι και προσεκλήθητε στην τελευταία συνεδρίαση και τα κρατή-μέλη ζήτησαν να δοθούν περισσότερη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων με κατεπήγοντα τρόπο και είπαμε ότι επήγει τέλο πάντων υπόθεση της Λιβύης και το καταπίστευμα ήταν ένα βασικό εργαλείο για να βοηθηθεί και η κατάσταση και έτσι να έχουμε την επανένταξη των μεταναστών που ήταν στις ε, φυλακές να πάνε στις κοινότητες βάσεις με αυθεντικά αναπτυξιακά προγράμματα. Δεν γίνεται έτσι στο γόνατο η ένταξη. Χρειάζεται πλαισίωση, χρειάζεται κατάρτιση και τελικά υποστήριξη ε, στην κοινότητα βάση του. Να τι θα πει ανάπτυξη. Και το άλλο θέμα που έχει σχέση με τις ε, ΜΚΟ 22% από το καταπίστευμα πάνε με συμβάσεις ε, στις ΜΚΟ 43% στο 5% ε, στις κυβερνήσεις και 30% πάνε σε διεθνείς ε, φορείς διεθνείς οργανισμούς τα κρατεί μελη και οι φορείς τους η FD και λοιπά και όπως και το OEM καλύπτονται μέρη από το καταπίστευμα οπότε τελικά το 50% του καταπιστεύματος ε, πάνε στις διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ. Ε, επίσης να σας πω για την αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στα διαχειριστικά όργανα. Αυτό όμως δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Αυτό είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Για τον Ήγερο τώρα, κάτι που είπατε όσον αφορά την διάλυση των ε, δικτύων των δουλεμπόρων των ε, διακινητών πλήση του τον εκεί και η κυβέρνηση της χώρας ήρθε να σας συναντήσει και να συζητηθεί το θέμα και εμείς πλησιώσαμε, βοηθήσαμε στην διάλυση των δικτύων την κυβέρνηση. Και τρέχουμε κάποια προγράμματα για τον πληθυσμό, τόσο ώστε να υπάρχουν εναλλακτικέ για να είμαστε ειλικρινεί, ε, ένα αλλακτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ποτέ δεν θα έχει τι ίδιε οικονομικές ευκαιρίες για τον κόσμο γιατί πολύ περισσότερα βγάζει ένας κτηνοτρόφι ή από ένα κτηνοτρόφι ή ένα γεωργό. Επομένως υπάρχει δυσκολία υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων αλλά εμεί προ τα εκεί πασχίζουμε. Και για να ολοκληρώσω Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τις τοπικές αρχές. Έχουμε διπουργικές συναντήσεις στην ε, Μπουρκίνα Φάσο για το καταπίστευμα και με άλλες χώρες και εκπροσωπούνται οι εμπλεκομένες χώρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Καταπιστεύματος και στην ε, Επιχειρησιακή Επιτροπή. Επομένως, είναι αβάσιμες οι σχετικές ε, επικρίσεις όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής, της στρατηγικής του καταπιστεύματος τώρα για όσα προγράμματα εξελίσσονται επί τόπου, ε, έχουμε συντονισμό, έχουμε συμπληρωματικότητα και ε, το καταπίστευμα ασχολείται με την καταπολέμηση της φτώχειας, με την καλή διακυβέρνηση τη αιτία της μετανάστευσης. Στη Δυτική Αφρική αυτά αποτελούν βασικό σκοπό της εταιρικής μας σχέσης. Έχουμε όλοι το ίδιο στόχο. Και θέλουμε να έχουμε τέτοιου είδου blending στην απασχόληση, στις υποδομές, στη γεωργία και γι' αυτό και θέλουμε έτσι να λειτουργούν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε που να υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις μακροπρόθεσμα επίσης. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα πρέπει να αρχίσω να σας ασκώ πίεση για να προχωρήσουμε. Δύο πράγματα θέλω να προσθέσω εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σας πω δύο λόγια για το εξής. Για το κατά πόσο η χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Ταμείου πηγαίνει και σε χώρες εκτός ΑΚΕ, σας απαντούμε όχι. Όχι, γιατί ε, δεν είναι επιλέξιμες. Από πλευράς Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού το βασικό εργαλείο που δίνει χρηματοδότηση στο φάκελο για τη Βόρεια Αφρική είναι το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για τη Γειτονία. Έχουμε και κάποια κονδύλια που έρχονται από το Εργαλείο Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΠΑΝΑΦ για την ε, Παναφρικανική Ήπειρο, αλλά όχι από το EDF, όχι από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Ε, επίσης, να απαντήσω στη βουλευτή που μας έδωσε το ερώτημα για τη Λιβύη. Είναι αληθές ότι έχουμε ένα πρόγραμμα για τη Λιβύη μεγάλο, άνω των 46 εκατομμυρίων, που μεταξύ άλλων ε, επωφελεί και την, Λιβύη, την λιμενοφυλακή, την ακτοφυλακή της Λιβύης. Όλοι ξέρουμε σε, ποιο, ε, σε πόσο δύσκολο πλαίσιο ζει η χώρα αυτή και έχει και τη μεγαλύτερη επιφάνεια διά, έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα της Μεσογείου από ότι ε, οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Έχουν σώσει 40.000 ανθρώπους μόνο πέρσι. Δεν είναι τέλειο το πρόγραμμά μας. Είναι ευάλωτη χώρα, αποτυχημένη χώρα αν θέλετε, έστω να την πούμε failed state, αλλά το πρόγραμμά μας στοχεύει να δώσουμε εκπαίδευση στη, στους λιμεδοφύλακες και στα μέλη της ακτοφυλακής και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, πολύ σύντομα, πολύ σύντομα παρακαλώ θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την απάντηση. Θέλω όμως να τονίσω το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να αξιολογήσει κανείς την ύπαρξη ε, της περιοχής διέρευνας και διάσωσης. Ακόμα και αν λένε οι αρχές της Λιβύης ότι έχουν τη μεγαλύτερη ζώνη έρευνας και διάσωσης και που το λένε προλίγο ας πούμε λίγων ημερών μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή με το μωρό της και μία άλλη γυναίκα εγκαταλείφθηκε με το μέσο της θαλάσσης μετά από παρέμβαση των αρχών της Λιβύης. Ε, δεν είναι δυνατόν να στηρίζει κανείς την ακτοφυλακή της Λιβύης γιατί δεν έχει αλλάξει καθόλου τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και η χρηματοδότησή μας το μόνο που κάνει είναι να τους αυτή την κατάσταση και αυτά που κάνουν εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι κάτι που λέει η που θα πρέπει να το εξετάσουν ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο διοίκησης. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και σημειώνω ότι Παρασκευή απόγευμα είναι δύσκολο να συνεδριάσουμε και να έχουμε παρουσίαση για να ασκήσουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο και ο διευθυντής από την αρμόδια γενική διεύθυνση θα πρέπει να το γνωρίζει. Και αν δεν έχουμε βουλευτές παρόντες, θα έχουμε μέλη της διοίκησης του Κοινοβουλίου παρόντα για να ελέγχουν το τι γίνεται. Επίτηδες, ε, δηλαδή, είναι δύσκολο που μεταθέσατε τη συνεδρίαση για την Παρασκευή απόγευμα γνωρίζοντας ότι ε, δυσκολευόμαστε και θα προχωρήσουμε στο σημείο 10. Θα είμαστε σύντομοι γιατί έχουμε πάρα πολλούς πρέσβεις από χώρες ΑΚΕ και έχουμε και το Γενικό Γραμματέα που περιμένει να συζητηθεί το κοτονού. Όμως είναι εξίσου σημαντικό να συζητήσουμε το σημείο 10 για τη δημιουργία του Ταμείου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Συνάδελφοι, είναι αυτό πολύ σημαντικό γιατί είναι το πρώτο από τα νομοθετικά μέτρα, τα νέα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μιλούμε για ένα εσωτερικό ταμείο μετανάστευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρηματοδοτεί κυρίω η Γενική Διεύθυνση Home Εσωτερικών. Με βάση το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο προπολογισμό αυτό να αυξηθεί 2,6 φορέ για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Δηλαδή να διπλασιαστεί συν άλλο τόσο. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να γίνουν και ε, έχουν σχέση με τις επιστροφές στη χώρα προέλευσης. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, εμεί προσπαθούμε να συνεισφέρουμε μέσω τη ε, γνωμοδότησή μα. Η ΑΦΕΤ επίση ε, θα καταρτήσει γνωμοδότηση. Επιτροπή επί τη ουσία, αρμόδια είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θα ψηφίσουμε στι 19 του Σεπτεμβρίου. Θα δώσω τώρα μέσω στο λόγο στην Έλλη Σλάιν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η αύξηση λοιπόν του προϋπολογισμού για το άσυλο και τη μετανάστευση είναι κάτι που οφείλουμε να καλωσορίσουμε. Είναι ένα θετικό βήμα προς ε, την δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης στην Ένωση. Το νέο Ταμείο λοιπόν Ασύλου και Μετανάστευσης μπορεί να συνεισφέρει εάν οι στόχοι του ε, τεθούν με σαφήνεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ε, μεταναστών, να βελτιώσουν τις συνθήκες ε, υποδοχής και τις ε, συνθήκες ε, ασύλου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρομερές ελλείψεις και αυτό είναι η αιτία του χάους που παρατηρούμε στη διαδικασία ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται πως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις επιστροφές και το ρόλο που θα παίξει το Ταμείο Ασύλου στην εξωτερική και όχι στην εσωτερική διάσταση. Τα θέματα που μόλις συζητήσαμε, το καταπίστευμα για την Αφρική ας πούμε κτλ ε, θα ε, είναι πολύ σημαντικά ως μέρος του ε, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίστη ότι η κατανομή των κονδυλίων θα γίνεται υπό προϋποθέσεις και τα ποσά αυτά δεν θα ε, διατίθενται για να ε, δίνουν κίνητρο για επιστροφές ή ανα, ε, αναγκαστικές επιστροφές. Αυτό μου φαίνεται πως αναφέρει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης χρειάζεται να φροντίσουμε για να υπάρχει συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο σχετικά με το άσυλο. Ε, προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην ε, γενικότερη ε, χωρητικότητα και στις χώρες προέλευσης. Επίσης, οι εθελοντικές επιστροφές θα πρέπει να συνοδεύονται και από μεσό και μάκρο πρόθεσμα μέτρα προς όφελος των ευάλωτων ομάδων μεταναστών. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, ιδιαίτερα τα παιδιά και να παρέχετε φροντίδα και σε πόρη για αυτές. Χρειάζεται επίσης προώθηση νομίμων οδών μετανάστευσης, ε, νέων θεωρήσεων για παράδειγμα εισόδου και ε, σε γενικές γραμμές νομίμων διάβλων. Αυτή η νόμιμη διάβλη είναι η μεγαλύτερη έλλειψη που αντιμετωπίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική ασύλου και η δημιουργία λοιπόν νόμιμων διάβλων είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την εμπορία ανθρώπων και να σώσουμε ζωές στη θάλασσα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ένας μόνιμος διάλογος και ε, μηχανισμός παρακολούθησης και ελέγχου που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε την εφαρμογή ε, και την υλοποίηση των κονδυλίων. Ας εστιάσουμε επίσης και σε ορισμένα θετικά στοιχεία του νέου μέσου. Σίγουρα δεν είναι λίγα, όμως αυτό που με ανησυχεί είναι ότι γίνεται λιγότερη μία στο άσυλο και σε αυτά που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να φροντίσουμε ότι τα χρήματα θα δετίθεται προς τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου και ε, πώς ε, όλοι θα ε, απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα όπως προβλέπει και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βλέπουμε ότι 30% ε, των χρημάτων πηγαίνει στο άσυλο, 40% στην μετανάστευση και άλλο ένα 40% στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ δημιουργούνται κίνητρα για τα κράτη-μέλη ε, έτσι ώστε να ε, εστιάσουν περισσότερο στην επιστροφή, στην καταπολέμηση της ε, μετανάστευσης και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε και χρειάζεται συζήτηση. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Αυτή είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να γίνει μια γενική παρουσίαση ε, κύριε Χιμένεθ και κύριε Κέγγε έχουν ζητήσει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τη συνάδελφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέγονται τώρα που δημιουργείται αυτό το νέο ταμείο. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να είμαστε σκιώδεις εισηγητές. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή του και βεβαίως να δούμε ποιο, πόσα χρήματα πηγαίνουν για το, ένα, για το ένα σκέλος και πόσα για, για το άλλο. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε στην ίδια βάρκα, ούτε να αξιοποιήσουμε τη μεταναστευτική πολιτική για να καταφερθούμε εναντίον της Ευρώπης. Στις χώρες μας και στην Ιταλία ξέρετε πώς έχουν αξιοποιηθεί όλα αυτά. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αυτός πιο ανθρωπιστής από τον άλλον. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ε, περισσότερο θύμα από τον άλλον και ότι ο άλλος δεν είναι. Όσοι έρχονται από τη Θέουτα θεωρούνται ε, εγκληματική οργάνωση που είναι θύλακος ισπανικός στη Βόρεια Αφρική και ε, τα αντίθετα έλεγαν ε, άνθρωποι του κόμματός σας όταν ήταν αυτοί στην εξουσία. Δηλαδή, ε, οποιοδήποτε κόμμα είναι γελίο να αξιοποιεί τη μετανάστευση για να παίξει πολιτικά παιχνίδια και πολιτικές σκοπιμότητες. Ε, δεν, το ίδιο γινόταν και με τα ναρκωτικά στην ε, Λατινική Αμερική και στην Κεντρική Αμερική. Δεν έχει σχέση ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα και φαινόμενα ως εργαλείο για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Πρέπει να δουλέψουμε από κοινού και να βοηθήσουμε τα σύνορα, θα το ζητήσουν οι χώρες μας και μάλιστα επισταμένως. Οι κυβερνήσεις είναι αριστερές και στη δική μου περιοχή και θα το ζητήσουν αυτό. Είναι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα στη ρίζα του. και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και ελπίζω ότι θα γίνει μια έκθεση ε, που θα μας ενώνει όλους. Συμφωνώ απολύτως. γιατί αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να εξαλείψουμε το φαινόμενο στη ρίζα τους, να μην έρχονται, γιατί αν δεν έχουν δουλειά εκεί θα διασχίσουν τα 16 χιλιόμετρα και είναι τεράστια μπίζνα αυτή. Το ξέρουν ήδη από πριν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις πότε θα φύγει μία βάρκα, ένα λαθρεμπορικό, πότε θα σαλπάρει. Το ξέρουν από πριν. Όλοι το ξέρουν. Και πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη. Ούτε με να μ' αρέσουν οι επιστροφές. Και ούτε όλα τα κράτη με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι δημοκρατίες, δυστυχώς. Αλλά με αυτούς έχουμε να κάνουμε και πρέπει να έχουμε ρεαλιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Η Σεσίλ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ λέει κυρία Κέγγε. Και εγώ να σας πω τη γνώμη μου για την συγκρότηση, για τη δημιουργία αυτού του ταμείου. Με προσοχή που παρακολουθώ τις εξελίξεις είναι σαφές ότι δεν υπάρχει μία και μόνη λύση για να μπορέσουμε να ε, ανταμοκριθούμε σε αυτή την μαζική κινητοποίηση που ονομάζεται μετανάστευση και αν έχουμε αφετηρία την ιδέα ότι δεν μπορούμε να φρενάρουμε την μετανάστευση ε, ε, ε, προσοχή, μην, ξεκινήσουμε σε λάθος βάση. Είναι ιστορικό, είναι φαινόμενο αιώνων. Κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Κινείται, μετακινείται ο κόσμος και οπότε απλώς θα πρέπει να δούμε για το πώς θα διευκολύνουμε τη ζωή αυτών που προσπαθούν να μετακινηθούν ή θα πρέπει κάτι να κάνουμε για τις υποκείμενες αιτίε. Δεν είναι δυνατόν να τους ε, φρενάρουμε, να τους κλείσουμε στο, στο χωριό τους. Θα πρέπει επομένω ε, παντού και στον Νότο και στον ε, Βορρά να ισχύσει αυτό. Γιατί δεν θα πρέπει να διαφοροποιούμαστε μεταξύ κάποιου ε, που προέρχεται από συγκεκριμένο μέρος του πλανήτη και να, να του πούμε ότι μπορεί να ταξιδέψει μόνο σε δύο χώρες και ένας που έρχεται από ένα άλλο μέρος του πλανήτη να μπορεί να ταξιδέψει σε 150 χώρες. Άρα θα πρέπει να δούμε ότι ό,τι επιστρατεύσουμε θα πρέπει να κατατείνει ή στο να διευκολύνει τη ζωή όλων αυτών των ε, ανθρώπων. Και ε, τελικά ο στόχος θα πρέπει να είναι εξασφάλιση ευημερίας για όλους τον ε, πλανήτη. Όχι, δεν είναι αυτό μια ουτοπία. Αν εμείς δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση, ε, τότε αρχίζουν ε, οι προτάσεις, οι λύσεις ε, που έχουν σχέση με ασφάλεια, οι επαναπροωθήσεις. Η Αφρική έχει πόρους, είναι πολύ πλούσια και θα πρέπει να μπορεί να ωφελεί στον κόσμο με αυτούς τους πόρους. Πριν αυτοί έρθουν εδώ, να αποφύγουμε την λαϊκιστική λογική. Να δούμε το πώς οι πρώτες ε, ύλες δεν θα ληστεύονται για τα τηλέφωνά μας και όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι πρόκειται για ε, μετακινήσεις που φέρνουν κόσμο που περισσεύει από την δική μας ε, επικράτεια. Θα πρέπει επομένως να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την υπόθεση αυτών όλων των ε, προσώπων και να δούμε τι θα γίνει σε όλες τις φάσεις από την ε, προέλευση, την διαμετακόμιση μέχρι την ε, άφηξη. Αν είναι να κάνουμε κάτι στην χώρα προέλευσης θα πρέπει να λαμβάνει την αξιοπρέπεια γιατί η προσωπική ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι η πρώτη προτεραιότητα. Να μην θεωρούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι ε, και ότι οι έσχατοι και δεν μπορούν να μείνουν στη χώρα μας. Έχουμε ένα σωρό διεθνείς συμφωνίες, ας τις στηρίσουμε. Και με αυτό θα κλείσω. Εδώ το κοινοβούλιο είναι βήμα δημοκρατίας. Πρεσβεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ας τα υλοποιήσουμε και να δούμε μήπως με αυτό το ταμείο μπορούμε κάτι να κάνουμε σε κάθε φάση του μεταναστευτικού φαινομένου. άλλη έχουμε το κοντινό που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πρόκειται να συζητηθεί. Στην συνέχεια, κύριε Σαφχάζος, θέλετε το λόγο γιατί πρόκειται για απλώς για μια πρώτη συζήτηση. Σαφχάζος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα, κυρία Πρόεδρε, θα εκφράσω την ε, προσωπική μου άποψη. Δεν θα σταματήσουμε τη μετανάστευση χωρίς να αναπτύξουμε την Αφρική, χωρίς να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε. Η Αφρική στους Αφρικανούς πρέπει να ανήκει και έχει τεράστιες δυνατότητες αυτό το πράγμα και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το 2050 ο πληθυσμό τη Αφρική θα είναι αυξημένο κατά ένα δι. Ό,τι και να κάνουμε, δεν θα σταματήσουμε αυτέ τι ροέ. Επομένω, δεν θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε και να ελέγξουμε αυτές τις πυροές παρά μόνο εάν αναπτύξουμε ε, την Αφρική. Και αυτό είναι το δεύτερο μέρος της παρέμβασής μου. Από τη μία πλευρά, το ελεύθερο εμπόριο, το γεγονός ότι έχουν ανοίξει αγορές των πρώτων υλών σε όλες τις εταιρείες. Το γεγονός ότι ε, είναι όλοι αντίθετοι στις κρατικοποιήσεις και στην κατανομή του πλούτου για την ανάπτυξη της Αφρικής. Όπως λέω εγώ, η Αφρική ανήκει στους Αφρικανούς. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στην φτωχοποίηση των χωρών και στην αποσταθεροποίηση. Οι παρεμβάσεις μας στην ε, λαϊκή δημοκρατία στο Κονγκό, η Δύση παρενέβη εκεί και στο Κονγκό και στη Συρία και στη Λιβύη και αλλού. Ε, η Συρία ίσω να αφαιθεί κατά μέρο γιατί δεν έχουν τελειώσει εκεί τα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρουμε ότι η Δύση έχει παρέμβει στι αιστείε τη αποσταθεροποίηση. Και αν μπορούσαμε να σταματήσουμε τι ροέ με τα σύνορα, θα, θα είχε γίνει. Μπορεί εγώ να είμαι πιο πολύ υπέρ της αποτελεσματικότητας των εθνικών συνόρων. Παρ' όλα αυτά και να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης θα παραμείνει το πρόβλημα. Θα ήθελα να καταγγείλω κάτι που είναι πραγματικότητα και το είδα και στο κοσυφοπαίδιο. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει συμμαχούν με τι διάφορε μαφίε. Υπάρχουν πολύ γνωστέ μη κυβερνητικέ οργανώσει που έχουν συνδεθεί και με οργανώσει που ασχολούνται με εμπόρια ανθρωπίνων ειδών και εμπόριο οργάνων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταγγείλουμε. Και δεν υποφέρω ε, πίσω από το ανθρωπιστικό σκέλος τελικά να κρύβεται το οργανωμένο έγκλημα. Ναι, το οργανωμένο έγκλημα και το ε, επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άρης Βαλίλα από τη Γενική Διεύθυνση Χόμαν, προφέρω σωστά το όνομά σας. Να είστε ε, πολύ σύντομος παρακαλώ. Ξέρω πόσο σας έχω κάνει να περιμένετε, αλλά είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε. Αν έχετε κάτι να προσθέσετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Τα σημειώνω. Ε, γνωρίζετε ότι αυτή είναι η έναρξη της διαδικασίας. Οριστικοποιήσαμε τις προτάσεις που ξεκίνησαν το Συμβούλιο, ξεκινήσαμε τις παρουσιάσεις στο ε, ε, Συμβούλιο. Συζητούμε πολλά για την κατανομή των κονδυλίων Το 5% δώσαμε μόνο μπροστά, 10% για την ενδιάμεση αξιολόγηση. Είναι πολύ δύσκολο να αναθεωρηθούν εκ των υστέρων οι, ο τρόπος με τον οποίο έχουν μοιραστεί τα χρήματα και στις αξιολογήσεις μας είχαν πει ότι η ευελιξία είναι πολύ σημαντική. Επομένως, γι' αυτό αυξήσαμε την ευελιξία και δώσαμε μεγάλο προσωστό μπροστά. Το 10% έχει τεθεί κατά μέρος για την ενδιάμεση αναθεώρηση, το 40% ε, έχει τεθεί κατά μέρος για το thematic facility εργαλείο για θεματικές ενότητες που θα δίνονται αυτά τα ε, χρήματα καθ' όλη τη διάρκεια δράσης του προγράμματος για διάφορες θεματικές ενότητες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του να έχουν αναθεωρηθεί κάποια στιγμή προτεραιότητες, να έχουν αναθεωρηθεί οι στόχοι. Στην αξιολόγηση επίσης μας είπαν ότι το σημερινό και εφιστάμενο πεδίο εφαρμογής είναι μια χαρά. Αυξήσαμε την ευελιξία μας, αυξήσαμε τα επίπεδα χρηματοδότησης. Το είπε και η κυρία Ντάλη αυτό. Μένει να δούμε την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Άσυλο και ενσωμάτωση 30% ε, των κοδηλίων. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να μην προχωρήσουμε γιατί θα συντάσετε την έκτασή σας για αρκετό καιρό. Είναι μια πρώτη προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η συγγήτρια, για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Περιμένω να συνεργαστώ και με τους λοιπούς συναδέλφους. Είναι πολύ θετικό να ε, δουλέψουμε μαζί για να καταλήξει η Επιτροπή μας σε μια ισχυρή θέση με τη γνωμοδότησή της. Θα δούμε ποια είναι τα θέματα που μας ανησυχούν, κάποιες ελάχιστες ε, ε, κατανομές κονδυλίων για, για την παράτυπη μετανάστευση, να φανεί η διαφορά μεταξύ της εξωτερικής δαπάνης και της εσωτερικής δαπάνης, να φανούν οι νέες διαχωριστικές ε, γραμμές μεταξύ του νέου ESF ε, Plus και του εργαλείου του προηγούμενου. Δεν είναι πολύ σαφή όλα αυτά ακόμα. Να μην γενικεύουμε όμως ότι όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, συνεργάζονται με τις μαφίες. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με αυτές. Και στην Ιταλία έχουν υπάρξει τέτοιοι ισχυρισμοί που κατάπεσαν, κατέρευσαν. Ξέρω ότι η περίπτωση για την οποία μιλήσατε. Οι κατηγορίες αυτές ε, δεν έστεκαν και οι Ιταλικές αρχές τελικά τις απέσυραν. Είναι πολύ δύσκολο να γενικεύει κανείς. Πράγματι πρέπει να ενισχύσουμε το μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογωμένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη θα υπάρξουν στο μέλλον πολλές ευκαιρίες έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να συζητήσουμε την έκθεση και όλα αυτά που μας απασχολούν. Περνάμε τώρα στο σημείο 11, τη μελλοντική συμφωνία Κοτονού. Ιδιαίτερα την διαπραγματευτική εντολή για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ε, ΑΚΕ. Δεν είναι πρώτη φορά που Συζητάμε το θέμα αυτό. Στο Κοινοβούλιο έχουν εγκριθεί ψηφίσματα για το μέλλον της Συμφωνίας Κοτονού. Ο Νόρμπερτ Νόιζερ είναι ο εισηγητής και είναι εδώ. Νομίζω όμως πως είναι η πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα αυτό από τη στιγμή που εγκρίθηκε η διαπραγματευτική εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για να δούμε τι έχει προκύψει στο μεταξύ. Έχουμε μαζί μας τον Πάτρικ Γκόμες, Γενικό Γραμματέα ε, για τις χώρες ΑΚΕ, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τη διαπραγματευτική εντολή. Επίσης, να καλωσορίσω τους πρέσβεις, ε, επιτελείο πρεσβειών από τις χώρες ΑΚΕ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπουμε λοιπόν σε καλή συνεργασία μαζί σας τους ερχόμενους μήνες. Θα δώσω τώρα το λόγο σε εσάς τον ε, Κουν Ντούνς που τον γνωρίζετε ίσως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπο της ΕΕΔ. Κύριε Κουν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πράγματι να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής. Πιστεύω πως είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, διότι τώρα μπαίνουμε σε μια νέα ε, περίοδο μετά την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής. Τώρα τόσο η πλευρά της Ένωσης όσο και η πλευρά των χωρών και έχουν τη διαπραγματευτική εντολή. Ε, επίσημα λοιπόν έχει γίνει η έναρξη των διαπραγματεύσεων μέσω ανταλλαγή επιστολών ε, ανάμεσα στον Επίτροπο Μίμητσα και τον Γενικό Γραμματέα Μπιαγκόνε ε, των χωρών ΑΚΕ. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν και επίσημα οι διαπραγματεύσει και αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσει να είναι ισχυρή η δέσμευσή μας γιατί αυτό θα καθορίσει και την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζετε, ο Επίτροπο Μίμητσα παρουσίασε το περιεχόμενο των ε, συστάσεων στην Επιτροπή ανάπτυξη ήδη τον Ιανουάριο. Μετά την έγκριση των αποφάσεων του Συμβουλίου τον Ιούνιο έχουμε ε, συγκεκριμένες ε, οδηγίες για τι διαπραγματεύσει που μοιάζουν λίγο πολύ με τις συστάσεις που έχουμε παρουσιάσει και συζητήσει μαζί σας. Και τώρα έχουμε λοιπόν την οριστική διαπραγματευτική εντολή που αφορά την διερθρωτική ε, συμφωνία ε, η οποία περιέχει τρεις ε, ισχυρούς πυλώνες, είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία και σκοπό έχει μια απλουστευμένη θεσμική δομή που θα δίνει έμφαση στις ε, στρατηγικές προτεραιότητες που έχουμε εντοπίσει. Ε, και οφείλω να ομολογήσω ότι προσπαθήσαμε ε, πολύ καιρό με τα κράτη-μέλη να προσέξουμε την διατύπωση, να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες. Νομίζω όμως πως το τελικό αποτέλεσμα είναι αρκετά εξισορροπημένο. Και μάλιστα αν συγκρίνει κανείς τη διαπραγματευτική εντολή με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διαπιστώσει ότι πολλά ε, βασικά σημεία συμπίπτουν. Και αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συνεργασία των κρατών μελών. Και αναφέρομαι στην απαλυφή της φτώχειας, κυρίως το οποίο είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητά μας στη συνεργασία με τις ε, χώρες της Αφρικής, του Ειρηνικού και της Καραϊβικής. Και έπειτα ένα στοιχείο στη Συμφωνία του Κοτονού πολύ βασικό είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της μελλοντική μας συνεργασίας μετά το 2020. Τέλος, γίνεται έκκληση για ισχυρή ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο εξάλλου αναφέρεται και στο ψήφισμά σας. Θεωρώ, επομένως, ότι αν συγκρίνουμε την έκβαση των ε, συζητήσεων στο Συμβούλιο και αυτά που ε, αναφέρει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διαπιστώσουμε ότι το αποτέλεσμα είναι αρκετά, αρκετά καλό. Και φτάσαμε λοιπόν μετά από όλα αυτά στην ε, διαπραγματευτική εντολή. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου τον Κρίστιαν και εγώ θα επανέλθω αργότερα για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, Κουν. Θα είμαι λοιπόν και εγώ σύντομος. Με δύο λόγια, νομίζω πως δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι το πλαίσιο πολιτικής και οι προοπτικές της πολιτικής μια είναι παρόμοιες τόσο στο, στην εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην εντολή των χωρών ΑΚΕ. Υπάρχει το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε, το θεματολόγιο δηλαδή για μετά το 2020, η, στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης, Υπάρχει παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη. Υπάρχει συνένεση λοιπόν σε όλους αυτούς τους τομείς και έχουμε προσπαθήσει τόσο να ενσωματώσουμε τις πολιτικές μας για αυτούς τους τομείς όσο και να ε, προσπαθήσουμε να τις ε, μεταφέρουμε στην ε, συμφωνία μετά το Κοτονού. Γίνεται έντονη αναφορά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε πολλά σημεία. Σίγουρα υπάρχουν ατομικές διαφορές και μπορεί να αποτελέσουν ε, δυσκολία στις ε, διαπραγματεύσεις, όμως οι γενικές γραμμές ε, οι προτεραιότητε μας είναι οι ίδιες. Είναι βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι θέματα που είναι πολύ σημαντικά και για τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα η μετανάστευση ανθρώπινα δικαιώματα, διακυβέρνηση, κοινωνία των πολιτών. Αυτά είναι στοιχεία αρκετά εμφανής και στις δύο πλευρές και νομίζω πως ε, οι διαπραγματεύσεις θα είναι ενδιαφέρουσες. Προσπαθήσαμε λοιπόν στη δική μας διαπραγματευτική εντολή για την Αφρική, την Καρυβική και τον Ειρηνικό να ενσωματώσουμε τις προτεραιότητες που αναφέρονται ε, στο θεματολόγιο από τους εταίρους μας. Υπάρχει το θεματολόγιο για την Αφρική, υπάρχει κοινή στρατηγική με την Καραϊβική τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, σχετικά με τον ειρηνικό υπάρχουν τα αποτελέσματα του ε, φόρουμ των νήσων του ειρηνικού, του PIF, που μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τις επόμενες ε, εργασίες μας. Σίγουρα χρειάζεται να βρούμε κοινά σημεία στο, σε τομείς που αφορούν το μέλλον της, ε, και τη διάρθρωση της συνεργασίας μας και όχι τόσο στους τομείς πολιτικής. Η διαπραγματευτική εντολή ΑΚΕ βασίζεται έντονα στις υφιστάμενες δομές και προσπαθούμε να βρούμε μία δομή που, και μία μορφή που θα αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που έχουν λάβει η χώρα στην Αφρική, στον Ελληνικό και την Καραϊβική, διατηρώντας όμως τα ισχυρά θεμέλια που έχουν δημιουργηθεί από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Γνωρίζουμε επίσης ότι στην πλευρά των χωρών ΑΚΕ διεξάγονται ακόμα συζητήσεις, ιδιαίτερα στην ομάδα για την Αφρική, έτσι ώστε να μπορέσουν να ερμηνεύσουν με τον σωστότερο τρόπο ότι το τι θα σημαίνει για αυτούς η, μελλοντική, η δομή της μελλοντική συμφωνίας. Γι' αυτό και ο Επίτροπος Μίμητσα συμφώνησε να δοθεί μια παράταση ε, να ανασταλεί η, έναρξη, το, η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων έτσι ώστε η ομάδα της Αφρικής να ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις της. και να ενημερώσει τις, ε, τους υπόλοιπους εταίρους ΑΚΕ. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ε, με λεπτομέρειες ποια θα είναι η έκβαση των ε, διαβουλεύσεων αυτών, όμως γνωρίζουμε πως θα υπάρχει μια μεγαλύτερη και πιο έντονη διαφοροποίηση ε, στις διάφορες περιοχές και αυτό είναι ενδεικτικό των αλλαγών που έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. κατά τη διάρκεια δηλαδή ζωής της Συμφωνίας του Κοτονού. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι ο πιο έντονος ρόλος των περιφερειακών οργανισμών, κάτι που θα έχει άμεση σχέση με την ε, εφαρμογή της συμφωνίας στο μέλλον. Και επίσης, τα κράτη-μέλη επιθυμούν να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Και το πλαίσιο της εποχής μετά Κοτονού να συγχωνευτεί με τις υφιστάμενες δομές όπως για παράδειγμα την στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής ή Ευρωπαϊκής Ένωσης Καραϊβικής. Όπως είπα, γίνονται πολλές συζητήσεις ε, από την πλευρά της Αφρικής και μεταξύ Αφρικής και των υπόλοιπων εταίρων της Καραβικής και του Ειρηνικού. Ε, στις 14 Σεπτεμβρίου στην Αντίσα Μπέμπα η συνάντηση που θα λάβει η χώρα θα είναι καθοριστική σημασία για την ολοκλήρωση του διαλόγου με τις ε, χώρες εκεί, έτσι ώστε να εισέλθουμε και επίσημα σε διαπραγματεύσεις περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου το αργότερο. στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου νομίζω πως έχουμε ακολουθήσει και του, τις δικές σας ε, επιθυμίες να υπάρχει ένας ε, διάλογος για βασικούς τομείς πολιτικής πιο αποτελεσματικός από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να λαμβάνει χώρα σε τακτικά διαστήματα και να είναι προσαρμοσμένος ε, στις ιδιαίτερες περιστάσεις του κάθε εταίρου. Μπορούμε να το χωρίσουμε σε διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο χωρών, ε, ομάδων, περιφερειών, αλλά και ε, σε όλο το φάσμα των ε, χωρών και ο διάλογος επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται και από συνεργασία με άλλους φορείς, την κοινωνία των πολιτών, και την εσύσφυξη των σχέσεων τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των χωρών ΑΚΕ. Τέλος, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση και σε περιφερειακό όμως επίπεδο, με τις τρεις δηλαδή μεγάλες αυτές περιφέρειες, Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικό, προσπαθούμε ε, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ε, ρεαλιστική εικόνα της ε, πραγματικότητας. Και προσπαθούμε να δούμε πώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα καλύτερα στοιχεία των επιμέρους διαβουλεύσεων και ομάδων έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε συνολικό επίπεδο για να έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και Τώρα νομίζω πως ε, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να σας μιλήσει για τα επόμενα βήματα. Ναι, θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομος. Οι προτεραιότητες που έχουμε για το μέλλον είναι καταρχάς να βρούμε μια χρονική στιγμή, εκεί τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, για να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ένωση και στους ε, εταίρους των χωρών ΑΚΕ. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή. Ο Επίτροπος Μίμητσα, όπως ξέρετε, είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Ε, από την πλευρά των χωρών ΑΚΕ, ο Υπουργό Εξωτερικών ε, του Τόγκο, ο Ρόμπερτ Τουσέ, είναι επικεφαλή των διαπραγματεύσεων και αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να βρούμε την κατάλληλη χρονική στιγμή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Όπω είπα, τέλο Σεπτεμβρίου ή αρχέ Οκτωβρίου. Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα αφορά κυρίως ανταλλαγή απόψεων για τις προσδοκίες μας, τις στρατηγικές προτεραιότητες και των δύο εταίρων και την έβρεση κοινών σημείων για την δομή της μελλοντική συμφωνίας. Θα εξεταστούν επίσης πρακτικές πτυχές διοργάνωσης τόσο σε ό,τι αφορά τη δομή, όσο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. καθώς και διαπραγματεύσεις για τους ε, τοπικούς πυλώνες. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα και τον κύριο Γκόμες από την ε, πλευρά των Χρονακέ. Όπως είδατε, με χαρά μας ήρθαμε μαζικά εδώ κατόπιν της πρόσκλησής σας Μπράβο που το Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που στα σοβαρά είδε αυτή την περίοδο μετά την Κοτονού. Φτιάξετε αυτό το ψήφισμα ε, και αυτό θα πρέπει να είναι μια καινούργια αρχή και να δούμε τώρα ε, όλα αυτά που μας ε, ζητήσατε να σας πούμε για να δούμε τι θα γίνει με την πρώτη χρηματοδότηση αλλά τέλος πάντων οι χώρες ΑΚΕ Θέλω να υπάρχει μια εταιρική σχέση σφαιρική, συνολική, ολοκληρωμένη ενώ του 21ου αιώνα ε, και έτσι θα πρέπει να δούμε ε, το πόσο σημαντικά είναι τα στοιχεία του κεκτημένου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και όλα αυτά θέλω να δούμε τι γίνεται με τους στόχους μας, τι γίνεται με τις βασικές αρχές και επίσης για κάποια θέματα πάρα πολύ βασικά, οριζόντια, εγκάρσια τέλος πάντων και να δούμε τις στρατηγικές αυτές προτεραιότητας, να υπάρξουν οι συλλογματικότητες, να δούμε τι διαφορές υπάρχουν και έχουμε αυτούς τους θεματικούς πυλώνες και δίνουν την εντύπωση ότι είναι συντηρητικού χαρακτήρα. Όχι, το αντίθετο διαπιστώθηκε ότι είμαστε καινοτόμοι επί της ουσίας. Και ποια είναι η ουσία, αυτά που λέτε και εσείς στο κείμενό σας, στο ψήφισμά σας. Ότι έχουμε τώρα την ουσία του Δήματος, τον πυρήνα, τις στρατηγικές αυτές προτεραιότητες, τους στρατηγικούς αναπτυσιακούς στόχους. Αυτά θα πρέπει να κρατήσουμε. ότι αν θέλουμε όλες οι χώρες ΑΚΕ και οι 28, οι 27 τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν, θα πρέπει να δούμε πώς παγκόσμια θα συνεργαστούμε και πώς ε, αυτοί οι στόχοι θα διαπνέουν τις ε, σχέσεις μας. Πώς έτσι ε, θα έχουμε ως Ευαγγέλιο το κεκτημένο και έτσι αυτό να έχουμε ως ε, μπούσολα ε, είναι βέβαια ε, εγκάρσιο οριζόντιο θέμα η μετανάστευση. Κοιτούμε τι γίνεται με την κινητικότητα. Ε, με τέτοια θέματα μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να έχουμε ένα παγκόσμιο σύμφωνο ε, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν τώρα με κριτικό μάτι να δουν το φαινόμενο. Όπως ενωμένοι αντιμετωπίσαμε το θέμα της αλλαγής του κλίματος όσον αφορά αυτή την περίφημη συμμαχία ε, της φιλοδοξίας. Κοινή όχι, ο καθένας δίνει αλλού βέβαια το ειδικό βάρος και όπως είπατε και το λέει και η συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να χτυπήσουμε την φτώχεια. Η κρίζωσή της θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά και έχουμε τους πυλώνες ε, προς τούτο δεν πρόκειται απλώς για εμπόριο. Πρόκειται για υπηρεσίες, για εκβιομηχάνηση, για επενδύσεις. Ανταγωνιστικότητα μέσω του εμπορίου που να οδηγούν σε επενδύσεις και εκβιομηχάνηση. Άρα τέτοια δεν πρέπει να είναι η εμπορική συνεργασία. Δεν λέμε για απλή βοήθεια. 0,7-0,2% είπαμε ότι έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά θέλουμε μετακίνηση τεχνολογίας. Και έτσι, με τεχνολογική πρόοδο, να έχουμε μετασχηματισμό της οικονομίας μας και έτσι να χτυπήσουμε τη φτώχεια. Και πάμε τώρα στον τρίτο στρατηγικό πυλώνα, πολιτικός διάλογος. Και αυτό είναι οριζόντιο εγκάρσιο θέμα. Πολιτικά θέματα, βασικές αρχές, ανθρώπινα δικαιώματα, μετανάστευση. Και βέβαια εμφανίζεται ότι θα πρέπει να δούμε τις ε, αιτίες, τις ρίζες του φαινομένου. Δεν θέλουμε να ισχύσει η παλιά αρχιτεκτονική. Τώρα έχουμε νέα φάση στον 21ο αιώνα για την Κοτονού. Να λάβουμε υπόψη όλα όσα έχουν αναδειχθεί μέσω των οδηγιών. Να μην πούμε απλώς ότι χωρίς θεμέλια κάτι θα κάνουμε στις περιφέρειες. Ε, αυτό απονευρώνει την ιδέα. Είναι ένα χταπόδι χωρίς κεφάλια. Προσοχή επομένως, να μην απονευρώσουμε την πολιτική αυτή. Να υπάρξει θεμέλιο, βάση. Να υπάρξει συμπληρωματικότητα, επικουρικότητα, αναλογικότητα. Για αυτό και θεωρήσαμε ότι η ισομερής κοινοβουλευτική συνέλευση συνεργάζεται, βρίσκεται σε αρμονία με τις άλλες μας συναντήσεις. Άρα, προσοχή στην εκτεκτονική αυτή να έχει στέρεα θεμέλια. Τον Οκτώβριο. Αρχάς Οκτωβρίου θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδρομή να επικεντρωθούμε ακριβώς στη βάση στο θεμέλιο και έτσι να υπάρξουν αυτοί οι πυλώνες, αυτή η περιφερειακή συνεργασία. Αυτό να είναι ο πυρήνας, το επίκεντρο, να στηρίζονται σε βάση στέρεα. Για όλα αυτά τα οριζόντια θέματα τα οποία αναφέρθηκαν στο μνημονιό μας, αποτελεί ουσιαστικά μια σύνοψη της διαπραγματευτικής εντολής. Είναι κάτι σαν θέμα της σώτας των φύλων που θα πρέπει να διαπνεί κάθε πολιτική. Να, έχουμε αυτά τα 350 εκατομμύρια συνεργασία, ΑΚΕ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόκειται για κονδύλια του EDF, Αφρική, Ειρηνικός, Καραϊβική. Άρα, είναι διτό το διτή προσπάθεια, πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Βέβαια, είναι κοινή η βάση, αλλά έχει η κάθε περιφέρεια ρυθμίες. Α, πώς μιλούσαμε για τη Βραζιλία υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αυτά που λέει η Επιτροπή Στατικής Προτεραιότητας. Και όπως ε, τα το πετύχαμε με το κλίμα, να δούμε τι θα γίνει με την διαχείριση των ωκεανών, τι θα γίνει με την ρήπανση μόλυνσή τους. 16 στρατηγική ε, αναπτυξιακή στόχη Να γίνεται η χάραξη της στρατηγικής και να ακολουθεί το επιχειρησιακό κομμάτι και να δούμε πώς η θεσμική αρχιτεκτονική καλύπτει την πρόταση για τη χρηματοδότηση. Συμφωνούμε θα πρέπει να βρεθούν πόρε Λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια. Η διαχείριση του πυρήνα της προσπάθειας. Πάντα αυτό θέλαμε. Και θα μπουν στη διαπραγματεύσεις τα κράτη, τα, των κρατών και μάλλον, θα μπουν στην διαπραγμάτευση λαμβάνοντας υπόψη τι πόροι υπάρχουν. Να μην υπάρξει κατάτμιση αυτών. Λίγο στην Καραβική, λίγο νότιο τη Σαχάρα, λίγο σε Ασία Ελληνικό. Μα αν υπάρξει κατάτμιση τότε δεν έχουμε την απαραίτητη συνέπεια σε σχέση με τα όσα συμφωνήσαμε ως βάση, ω αφετηρία. Άρα ό,τι συμφωνήσαμε να αντικατοπτρίζεται στην συμφωνία. Και είχαμε το κείμενο του ε, εισηγητή, εγκρίθηκε. Οδηγούμεθα σε περισσότερη υποχρέωση λογοδοσία, σε περισσότερη διαφάνεια, ε, ισόφελος των πολιτών της Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα, πρέπει να έχει διαχρονικό χαρακτήρα. Αλλιώς δεν θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, κάποια δέσμευση κεφαλαίων που ισχύει σήμερα και όχι αύριο. Και δεν θα πρέπει να, ας πούμε, όπως με το Ιρανικό, με την κρίση αυτήν, ε, η άμυνα να αποκτά ξαφνικά προτεραιότητα αντί των άλλων θεμάτων όσον αφορά τον προπολογισμό. Γι' αυτό και ελπίζουμε αυτά να τα αλλάξουμε μετά τι επαφές με την Κομισιόν, γιατί προ το αυτά δεν αποτυπώνται σχετικέ οδηγίε. Εδώ να βάλω μια τελεία, γιατί έχουμε και άλλου που θέλουν τον λόγο. Έχουμε ε, τον πρέσβη από το Τόγκο για τις διαπραγματεύσεις σε υπουργικό επίπεδο. Ψηλούς, ε, ψόβαθμους διπλωματές από το Τσάδ. Υπάρχει μια ευκαιρία που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. All speakers. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση για τις και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται. Συμφωνείτε, λέτε και οι δύο, με τα του Κοινοβουλίου, όμως τις απόψεις σας ε, έχετε απόκληση μεταξύ σας και προσπαθώ να καταλάβω τι υπονοείτε και τι δεν λέγεται. Το σημαντικό είναι να δούμε ποια θα είναι τα βασικά ζητήματα που θα βρίσκονται στον πυρήνα των διαπραγματεύσεων. Βλέπω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση. Ε, δεν βλέπω εκεί κάτι. Ίσως ε, μπορεί να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν υπάρχει κάτι για την χρηματοδότηση και ποια είναι η παλιά συμφωνία, είναι, ποια είναι η διαφορά με την καινούρια. Ε, ποια στοιχεία απουσιάζουν, για να μπορέσουμε να τα μελετήσουμε όλα αυτά, πώς αλλάζει η εντολή η διαπραγματευτική και η εντολή μετά τη συμφωνία του Κοντονού. Σίγουρα έτσι θα διευκρινιστεί αυτή η γλώσσα για κατανόητη που έχουμε ακούσει ο Νόρμπερτ να κάνει την αποκωδικοποίηση της δύσκολης αυτής γλώσσας που ακούσαμε. Ευχαριστώ, Λίντα. Ευχαριστώ και τους ομιλητές σας. Ευχαριστώ και για τα κοπλιμέντα προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί ε, ξεκινήσαμε με το πρώτο θεσμικό όργανο, είμαστε το πρώτο θεσμικό όργανο, κάναμε τα μαθήματά μας ως κοινοβουλευτικοί, μελετήσαμε, δουλέψαμε, ε, μπορούμε να ασκήσουμε μεγάλη επιρροή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Καλό είναι βεβαίως και πολύ ωραίο να προσπαθεί κανείς να διαβάζει και να καταλαβαίνει και τα συμφραζόμενα και αυτά που παραλείπονται γιατί είναι ευκόλως εννοούμενα. Πετύχαμε πολλά θετικά. Αυτό είναι αληθές. Τώρα που ξεκινάει η νέα θητεία, η νέα διάρκεια ισχύω της Συμφωνίας του Κοτονού. Η καταπολέμηση της φτώχειας, η χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ισότητα των φύλων, η κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά περιλαμβάνονται και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Κάποια προβλήματα μένουν με τα εργαλεία που έχει αυτή η σύμπραξη χωρολακέ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινοβουλευτική τους διάσταση. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ κοντά στα συμπεράσματα των χωρών ΑΚΕ. Όσον αφορά το GBA. Στη ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν σε ορισμένες χώρες κάποιες, ε, κάποιοι ενδιασμοί γι' αυτό. Όμως οι διαπραγματευτικές οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος αναφέρουν ότι η συμφωνία θα ενισχύσει το, το κοινοβουλευτικό σκέλος στο περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο περιφερειακών εταίρων. Και άρα είναι εκτός ημερησίας διατάξεως η δημιουργία ενός μεγάλου GPA, ε, μιας ε, συνολικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Δεν είναι συντηρητική δομή το GPR, είναι κοινή, συνηθισμένη. Και μπορούμε να τις δώσουμε ένα νέο προφίλ, γιατί έχουμε νέους, νέες προκλήσεις να υψώνονται μπροστά μας. Επομένως είμαστε αρκετά κοντά στη θέση των χωρών ΑΚΕ και είμαστε κάπως ενάντια ε, στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Αυτό το ερώτημα είχα να θέσω για το μέλλον του GPA, τη συνολική συμφωνία Εταιρική Σχέσης και όχι μόνο στο επίπεδο περιφερειών, περιφερειακής εταιρική σχέσης, αλλά να υπάρχει και η παγκόσμια διάσταση. Πώς θέλουμε εμείς ως Ευρωπαίοι να απαντήσουμε σε αυτό το core management που ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, σε αυτή τη διαχείριση, αν θέλετε, από ένα πολύ βασικό κεντρικό πυρήνα. Θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, να συνεχίσουμε το διάλογο βεβαίως, Βλέποντας όμως το μέλλον, βλέπουμε ότι έχουμε χρόνο διαπραγμάτευσης περίπου για 1,5 έτος. Όμως σε ένα χρόνο θα λήξει τις εργασίες της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υφιστάμενη της ε, μορφή ε, μέχρι να έρθει καινούρια. Άρα, ε, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Να μας βοηθήσετε. Η ευχαριστώ. Ναι, είναι σημαντικό να έχουμε ορίζοντα συγκεκριμένο εν ώψη των κοινοβουλευτικών εκλογών, των ευρωεκλογών το Μάιο, τη σύσταση της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη συγκρότησή και του κ.ο.κ. Η Τερέσα Χιμένεθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω ισπανικά. Νομίζω ότι μια διαπραγματευτική εντολή για μελλοντική συμφωνία είναι πάντοτε μεγάλη ευκαιρία να βελτιώσουμε τα ήδη υφιστάμενα. Και εγώ είχα ρωτήσεις για τις ημερομηνίε και τις καταληκτικές προθεσμίες και με ανησυχεί η παρουσία του Μεξικού για, στις διαπραγματεύσεις για τον εξυγχρονισμό μιας συμφωνίας που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα έχουμε προβλήματα. Δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρουμε να κλείσουμε τη συμφωνία για λόγους ημερομηνιών και προθεσμιών. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ε, δέσουμε σφιχτά τη συμφωνία και να τα καταχειρώσουμε όλα αυτά. Τώρα, οι χώρες που είναι μέλη στο ΑΚΕ είναι πολλές και διαφορετικές. Έχουν διαφορετικούς πληθυσμούς, διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, διαφορετικό επίπεδο εισοδημάτων. Ποιες θα είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε με αυτή την τόσο μεγάλη ποικιλομορφία. Και σε σχέση με το στόχο 16 των ε, στόχων αναπτυξιακών της χιλιετίας. Μπορείτε να αναπτύξετε λίγο το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Πώς θα το κάνουμε αυτό από κοινού γιατί πρόκειται για μια παγκόσμια απειλή όχι μόνο στην Ευρώπη. Και άλλωστε στην Ευρώπη η τρομοκρατική απειλή είναι πολύ περιστασιακή σε σχέση με τις χώρες της Αφρικής όπου τα θύματα είναι πάρα πολλά ε, και είναι, ανήκουν στο γηγενή πληθυσμό από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Επίσης υπόθηκε ο τρίτος πυλώνας και το θέμα της μετανάστευσης και έχει υποθεί πανελειμμένος ότι οι χώρες ΑΚΕ θα πρέπει να εμπλακούν σε, αυτό το, ε, σε αυτή τη δράση. Ε, με ποια μορφή όμως μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Μαρή είναι η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Δεν ανήκω στην Επιτροπή σας, αλλά ασχολούμαι με τις ΑΚΕ και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σχολιάσω ε, το θέμα που εξετάζετε, τις χώρες ΑΚΕ δηλαδή. Έχει γίνει σημαντική δουλειά και θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας και εδώ εντό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση μεταξύ χωρών ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν προχωρήσει τα θέματα. Όλοι συγκλίνουν δηλαδή προς την ίδια κατεύθυνση, προς τον ίδιο στόχο και αυτό είναι πολύ θετικό. Έρχομαι στο ερώτημα που έθεσε ο Νόρμπερτ, ο συνάδελφος, για το μέλλον της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης. Είναι ένα σπάνιος τόπος, είναι ένα από τα σπάνια μέρη σήμερα όπου μπορεί κανείς να δουλέψει σε, με επίσημη μορφή, σε επίσημο πλαίσιο, ε, να μπορεί να εργαστεί μεταξύ Κοινοβουλίων Εθνικών, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κοινοβουλίων των χωρών του Καραϊβικής, της Αφρική, του Ειρηνικού κτλ. Σε αυτή τη διακοινοβουλευτική λοιπόν συνέλευση έχει γίνει πολλή δουλειά για να ανοίξουν νέοι δρόμοι και αυτό μας βοήθησε για να συντάξουμε τη Συμφωνία του Κοτονού. Και ε, οι χώρες ΑΚΕ μπόρεσαν να καταλήξουν σε κοινή θέση, τη λιγότερο αποκλίνουσα θέση σε σχέση με τους στόχους που αμφότεροι επιδιώκουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η κοινή διακοινοβουλευτική συνέλευση να παραμείνει, να μην εξαφανιστεί. Βεβαίως να βελτιώσει τη λειτουργία της, αλλά να διατηρηθεί να μην δουλέψουμε αποκλειστικά και μόνο στο περιφερειακό επίπεδο, γιατί τα θέματα και οι θεματικές ενότητες που μας απασχολούν, μας απασχολούν όλους εγκαρσίως. Τα απαντούμε και τα συναντούμε και προσκρούμε πάνω σε αυτά και στις χώρες της Αφρικής και στις χώρες Καραβικής και εδώ σε τα μας. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα. Άρα πρέπει να διατηρήσουμε μια διάσταση η οποία να μην είναι μόνο περιφερειακή. Αν σταθούμε μόνο στην περιφερειακή διάσταση θα έχουμε την τάση να διαιρούμε τους εταίρους μας και όχι να τους συνενώνουμε ε, πάνω σε ε, για θέματα που μας αφορούν. Αυτό καταρχάς είναι η πρώτη ανησυχία που ήθελα να εκφράσω. Δεύτερον, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόμαστε μια στρατηγική εταιρική σχέση με την Αφρική και ορισμένες φορές ακούω ανθρώπους από την Αφρικανική Ένωση να δηλώνουν και να λένε ότι θέλουν να φύγουν από τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο ΑΚΕ μετά τη Συμφωνία του Κοτονού και να δώσουν ε, έμφαση στη διμερή διαπραγμάτευση με τα δύο μέρη να είναι η Αφρική από τη μία πλευρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη. Η Αφρικανική Ένωση από τη μία, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη. Τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Έχουμε από τη μία στρατηγική κοτονού και νέα συμφωνία κοτονού και ένα σωρό δουλειέ εκεί και από την άλλη έχουμε στρατηγική που υπονομεύει την πρώτη μας επιδίωξη. Καταλαβαίνω και βλέπω τους προσανατολισμούς που αναδύονται μετά την πρώτη συμφωνία για το Κοτονού, όμως έχουμε και οικονομικές συνθήκες και σχέσεις προνομιούχες. Είναι σημαντικό λοιπόν να μιλήσουμε για την οικονομία ως παράγοντα ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει αυτό να το παραγνωρίσουμε ούτε να το παραμελήσουμε. Να απαιτήσουμε από την οικονομία να λειτουργήσει ως παράγοντας ανάπτυξης. Άρα να είναι μια οικονομία, οικονομική πολιτική που θα ασκείται για να καταπολεμήσει τις ανισότητες, την κλιματική αλλαγή, τη διαφθορά. Άρα να δώσουμε προτεραιότητα στο οικονομικό σκέλος και όχι τόσο στο ανεπτυξιακό, αλλά να το κάνουμε έχοντας τις δικλίδες ασφαλείας για να μην καταλήξουμε σε μια άγρια οικονομία ε, ε, που την έχουμε δει σε αφρικανικές χώρες και που καθόλου δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη. Άρα πρέπει να, έχουν παράγοντες, πρέπει να έχουμε παράγοντες ρύθμισης των αγορών έτσι όπως προβλέπονται και να προβλεφθούν αυτά στη νέα συμφωνία για το κοτονό. Ευχαριστώ η Μαρία παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τη δουλειά που έχετε κάνει και να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημοσίευση τη διαπραγματευτική εντολή. Ε, διότι με τον τρόπο αυτό έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ζητά το Κοινοβούλιο. Είναι πολύ ε, θετικό λοιπόν το ότι δημοσιεύτηκε η διαπραγματευτική εντολή και πετεύχθη η διαφάνεια. Σας ευχαριστώ και μπράβο σας. Έχω μια ερώτηση που αφορά τη μετανάστευση. Στη διαπραγματευτική εντολή αναφέρεται ρητά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαπραγμάτευση του άρθρου 13 θέλει ε, ενίσχυση ε, του σημείου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θέλει να κερδίσει το παιχνίδι της μετανάστευσης. Ε, αυτό συμβαίνει εδώ αναρωτιέμαι. Για μένα όμως ε, το ε, σημαντικό είναι το τίμημα το οποίο θα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Ε, ποιο είναι το τίμημα για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Συμφωνία με δικτατορικά καθεστώτα, συμφωνία με τον Ασάντα σου, με τις ε, ομάδες ανταρτών στην ε, Λιβύη. Ποιο είναι το τίμα που θα πληρώσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι που με απασχολεί υπό ποιες ε, συνθήκες και πώς θα επηρεάσει αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και άλλη μια ερώτηση. σε ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία. Στο κεφάλαιο 3 της διαπραγματευτικής εντολής του Συμβουλίου αναφέρεται γενικές γραμμές ε, μια ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες ΑΚΕ. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό ως ενίσχυση της συνεργασίας μέσω των ε, διεθνών ε, οργανισμών, με διεθνή φόρα. Ή κάνω λάθος. Εσείς, ε, ο κύριος Εγκόμες, έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα να μου δώσετε αυτής της ε, ενίσχυσης ε, της συνεργασίας. Να σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Φορολογική συνεργασία. Θα μπορούσε αυτό το θέμα να είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουν οι δύο και θα καταλήξουν σε κάποια κοινή αντιμετώπιση. Μετά. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο ακόμα σημεία. Η στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κύριος Γκόμες μας ε, ανέφερε το πόσο σημαντική είναι. Ερωτώ λοιπόν στην διαπραγματευτική εντολή αναφέρεται κάτι επί της ε, ουσίας για την ε, καταπολέμηση ε, των ε, προβλημάτων, ε, βρέσει λύσεων. Έτσι όπως το καταλαβαίνω όταν το διαβάζω, μου φαίνεται ότι δεν αλλάζει και κάτι. Δεν αναφέρομαι βέβαια στην γεωργική πολιτική, γιατί εκεί είναι λίγο πολύ καθιερωμένη και δρεωμένη πολιτική. Όμως σε άλλους τομείς υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, πώς θα δοθεί έμφαση στην αηφορία. Αυτό το καλοκαίρι που μόλις τελειώνει μας δείχνει πιστεύω ότι μας περιμένει στο μέλλον. Στην ε, Ευρώπη ειδικά ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα αυτά ε, και στις αγροτικές εκτάσεις στη χώρα μου, τη Γερμανία, τα λιβάδια ήταν καφέ, είχαν ξεραθεί τα πάντα. Υπάρχει λοιπόν κάποιο και πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση ε, της ε, κλιματικής για, και το πώς αυτό συνδέεται με τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλα τα κρατημέλη έχουν καταδείξει πως ε, θέλουν να δώσουν έμφαση στις εμπορικές συμφωνίες. Έχετε όμως ε, κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε ποιες είναι οι προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις χώρες ΑΚΕ. Μετά, αναφέρθηκε η δημιουργία, η επιθυμία μάλλον, για δημιουργία μιας ε, παναφρικανικής ε, εμπορικής ζώνης. Αυτό θα γίνει παράλληλα με τις ε, διαπραγματεύσεις διότι το θεωρώ σωστότερο να συνδυαστούν αυτές οι προσπάθειες, να μην γίνονται ξεχωριστά. Ε, και επίσης η κοινή διαχείριση των ε, πόρων ήταν κάτι που μέχρι τώρα λειτουργήσε λίγο πολύ σωστά. Ε, εσείς τι άποψη έχετε γι' αυτό, θέλετε αυτό να αλλάξει ή διαφωνείτε με το ότι έγινε σωστή διαχείριση από κοινού των πόρων. Αυτά προς το παρόν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Σεσίλη Κέγγε και μετά στους ε, πρέσβες εφόσον το επιθυμούν. Η κυρία Αζίζ ε, Μπαρούντ έχει ζητήσει το λόγο ε, πρέσβηρα του Τσάντ. Αλλά η κυρία Κέγγε έχει τώρα το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, Λίντα, με δύο ερωτήματα, τα οποία έχουν φυγεί και από τους προλέλησαντες. Πρώτα-πρώτα, το πρώτο το οποίο θέλω να πω για την ταξί είναι ακριβώς αυτό, όσον αφορά την αρχή αυτής της εντολής. Να δούμε πώς θα ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση, δηλαδή το μέλλον της ε, Ισομερούς Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕΕ. Και, θα ήθελα ε, να μου πούν το, το πώς σκέπτονται οι συνομιλητές μας όσον αφορά αυτήν ε, την ε, συνέλευση. Το πώς δεν θα την αναβαθμίσουμε και δεν θα ακολουθήσει ε, κάποιο είδους πισωγύρισμα. Για ένα σωρό λόγους θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση, αλλά όμως πρακτικά, τεχνοκρατικά, πώς το βλέπετε. Κάτι άλλο τώρα, όσον αφορά το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, πώς αυτό θα στριχτεί, τι είδους κίνηση θα γίνει για να υποστηριχθεί αυτή η νέα συμφωνία. Πεςτε μου τη γνώμη σε αυτά τα δύο σημεία. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Άζης Μπαρούτ που προεδρεύεται τη, του Επιτροπής των Πρέσβειων. Εσείς κύριε πρώτος, ναι, αφού το θέλετε. Να γιου Πλέντη. Προσπαθώ, προσπαθώ να διαβάσω ε, το γραφικό σας χαρακτήρα που φυσικά είναι καλύτερος από το δικό μου. Ε. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, μου δίνετε την ευκαιρία εδώ να τοποθετηθώ ενώπιον των βουλευτών. Για μας αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία για μας τις χώρες ε, ΑΚΕ να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε όσον αφορά την προκατευτική εντολή. Τι θα γίνει για αυτή την φάση κατόπιν της Κοτονού. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε είναι πάρα πολύ ενημερωτικά. Ό,τι ακούσαμε από όλους τον λόγο. Πρόκειται για την πρόταση της εντολής όπως παρουσιάστηκε από τον Γενικό Γραμματέα μαζί για τη διαχείριση των θεμάτων ΑΚΕ σας τα παρουσίασε όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Εντολή και όπως διαπιστώσατε δεν έχουμε κανένας είδους σημαντική διαφορά μεταξύ των εντολών. Η μόνη διαφορά υπάρχει όσον αφορά τη διάρθρωση, τη δομή των γράφων και έχουμε αυτές τις ε, ιδέες, τις προτάσεις, το θεματολόγιο για να μπορούμε να προχωρήσουμε και το πιο δύσκολο είναι και βλέπουμε με χαρά αυτά που είπε ο κ. Πούντα και θα τα συζητήσουμε όσον αφορά τη δομή αυτής της συμφωνίας, να δούμε πώς θα γίνει το χρονοδιάγραμμα, πώς τι θα γίνει με τους περιφερειακούς πυλώνες ε, κλπ. Ακριβώς σε αυτό το θεματολόγιο στο κάθε πλαίσιο. Δεν, υπάρχει εδώ πέρα θέμα απόκληση απόψεων, γιατί αυτό το θεματολόγια ένα προς ένα, θα τα εξετάσουμε και θα εξεταστούν τα τυχόν σημεία διαφωνίας. Και ως προεδρεύων αυτής της κεντρικής ομάδας που συγκροτήθηκε από τις χώρες ΑΚΕ θα σας πω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις με τους ε, Ευρωπαίους. Ακριβώς όπως είπε ο κύριος Γενικός έτοιμοι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ό,τι επιδέχεται βελτίωση. Θεματολόγιο, εγκάρσια ζητήματα, όλα αυτά τα οποία έχετε και στα δικά σας έγγραφα. Αυτά που μας παράσχουν την ε, επιβεβαίωση ότι υπάρχει καλή πίστη, καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Και δεν έχουμε κάποιο είδου διαφωνία. Και χαίρομαι για ένα ερώτημα που μας θέσατε. Και το ερώτημα που μπορεί να απαντήσει η Επιτροπή. Εμείς κάνουμε διαπραγματεύσεις σε αυτή την κοινή βάση που προτάθηκε από την Ευρώπη. Όλα αυτά καλύπτονται από την διαπραγματευτική εντολή μας. Όπως είπατε, χέρι-χέρι θα πάμε τέλος Σεπτεμβρίου για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Άντε, αρχές Οκτωβρίου. Πάλι σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή. Όπως είπαμε, έχει καινούριο ορισμό, η ευρωπαϊκή εντολή, εμείς τέλος πάντων δεν έχουμε πρόβλημα τη δική μας. Θα είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά πάνω από 40 χρόνια έχουμε εταιρική σχέση. Οπότε θεωρούμε ότι τα πράγματα θα έχουν αίσια εξέλιξη. Η Πρόεδρος. Κύριε, κύριε Ζησμπαρούτ, έχετε εσείς τον λόγο από το Τσάδ. Χαιρετίζω την Ομίγυρη και νομίζω ότι είναι τώρα μια ευκαιρία για να μιλήσουμε για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα και να έχουμε μια φιλική ανταλλαγή απόψεων. Και από αυτόν τώρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα πρέπει να προσθέσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Έχουμε την εντολή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ακριβώς που υπάρχουν κάποια στοιχεία. Πού χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση. Μιλούμε για την περίοδο μετά το κοτονού. Μιλούμε για συνεργασία που κάτσε 40 χρόνια και τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε εξελίξεις, είχαμε αλλαγές γεωστατικικές περιβαλλοντικές και άλλες. Και άλλες. Και έτσι αυτές οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να προετοιμάσουν το μέλλον που δεν είναι γεμάτο προκλήσεις. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αναφέρθηκε το θέμα του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε το μοναταστευτικό, όλα αυτά είναι οριζόντιο χαρακτήρα θέματα. Όλα αυτά μας απασχολούν όλους. Ε, είναι κοινή προσπάθεια. Θα πρέπει με προσοχή να τα αντιμετωπίζουμε. Είναι θέμα ηθικής υποχρέωσης πώς όλα αυτά θα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Όσον αφορά τώρα τους περιφερειακούς πυλώνες, δεν μπορούμε να μην λαμβάνει υπόψη ότι οποιαδήποτε περιφέρεια ή περιοχή έχει γνωρίσει κάποιες εξελίξεις, κάποιες ιδιορυθμίες που θα πρέπει έτσι να ειδωθούν. Και πιο σημαντικό όμως είναι το θέμα των κοινών ζητημάτων, των οριζοντίων θεμάτων που αντιμετωπίζονται βουλευτικά, Ε, αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και με τις επίσημες συνομιλίες να βρεθούν οι απαντήσεις. Που πρέπει τώρα όσον αφορά τις φιλοδοξίες της Αφρικανικής Ένωσης Θα χρειαστούν κάποιες διευκρινήσεις. Θα προχωρήσουμε τον Σεπτέμβριο προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν έχουμε περιθώρια για να κάνουμε λάθος. Δεν θα πρέπει να είναι κατατμημένες οι προσπαθίες μας. Ούτε μπορούμε να έχουμε κατά νου μόνο την περιφερειακή διάσταση. Πολύ σημαντικό το κεκτημένο ε, θα πρέπει με το κεκτημένο ως βάση να προχωρήσουμε. Μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτή η συνάντηση στην ε, Αφρικανική Ένωση. Ήδη έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις. Και βέβαια θα πρέπει να κυριαρχήσει η ιδέα της ενίσχυσης της, ε, του, του κριτηρίου των τοπικών, των περιφερειακών ρυθμιών Ό,τι κάναμε αυτά τα 40 χρόνια δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε ή να το αγνοήσουμε. Κάποιος μίλησε για συγκεκριμένη αντιμετώπιση Στι αναπτυσσόμενε χώρε ισχύει αυτό, ισχύει για ε, του στόχου ε, τη ανάπτυξη, ισχύει για τι χώρε ε, τη ε, ΑΚΕ, για τι διεθνεί συνθήκε. Και έτσι θα πρέπει να δούμε. Και εμείς πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτόν τον προβληματισμό των Ευρωπαίων εταίρων μας ε, και κυρίως των ε, Ευρωβουλευτών, γιατί πάντα λέγω ότι η προσπάθειά μας αρχίζει και τελειώνει με εκείνους. Οπότε θα προχωρήσουμε στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Οι διερμηνείς μας έχουν δώσει 10 ακόμα λεπτά. αλλά δεν χρειάζεται και να τα εξαντλήσουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Με λένε Μωαμέτη Γκέ. Ανήκω στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Παναφρικανικής Ένωσης εδώ στις Βρυξέλλες και παίρνω το λόγο για να σας πω το εξής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα του, της συμφωνίας μετά το Κοτονού για την Αφρικανική Ένωση, γιατί η συμφωνία θα δεσμεύσει την Αφρικανική Υπήρο στη συνεργασία της με την Ευρώπη, που παραμένει βασικός εταίρος της Αφρικής. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αυτών των συμφωνιών. Μία συμφωνία μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είναι συγκεκριμένη και να δώσει αυτά αποτελέσματα στους πολίτες αμφωτέρων πύρων. Σήμερα λοιπόν, στη συνεργασία αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιοι τομείς που συζητούνται σε φόρουμ εκτός Αφρικανικής Ένωσης. Θα συμφωνήσετε λοιπόν ότι όταν υπάρχουν παράλληλες διαδικασίες και διεργασίες, ουσιαστικά υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της δουλειάς όλων μας. Και γι' αυτό εμείς ε, δουλεύουμε για να έχουμε μια κοινή θέση ε, για την στάση και την ε, επιδιώξει μας για την Ευρώπη μετά το 2020. Στο Κικάλι λήφθη σχετική απόφαση και οριστικοποιείται η κοινή μας θέση. Το 1η Ιουλίου, στη 31η συνεδρίαση της ε, ε, Αφρικανικής Ένωσης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, συζήτησαν επί το θέμα αυτό και ανέθεσαν στο πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης να απευθυνθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αναβληθεί η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία του Κοτονού πριν μέχρι ότου ε, καταλήξουμε σε κοινή θέση ως Αφρικανική Ένωση. Στην Αντίσα Μπέμπα σε δύο εβδομάδες θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Εκτελεστικού της Αφρικανικής Ένωσης Δηλαδή, οι Αφρικανοί Υπουργοί Εξωτερικών ε, θα συνεδριάσουν, θα υπάρχει διευρυμένη συνεδρίαση με παρουσία υπουργών επιφορτισμένων με τα θέματα ΑΚΕ και η εντολή είναι να οριστικοποιήσουν την κοινή θέση των ε, χωρών της Αφρικανικής Ένωσης που θα είναι και η κοινή οριστική θέση της Αφρικής και μπορούν έτσι να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για τη συνεργασία μεταξύ των δύο υπήρων για την περίοδο μετά το 2020. Σας ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Ε, περιμένουμε τις εξελίξεις από τη συνεδρίασή σα το Σεπτέμβριο σε δύο εβδομάδες. Στον Κριστιαν και στον Πατρίκ να δώσω το λόγο για τα τελικά σχόλια. Τρία λεπτά ο καθένας μέγιστο. Κουν παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Λίντα και σας ευχαριστώ όλους. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά ξεκινώ με το θέμα που θέσατε εσείς. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα και αυτό προέκυψε. Πρώτον, η δομή της συμφωνίας. Ό,τι μπαίνει στους γεωγραφικούς πυλώνες μπαίνει εκεί και ό,τι δεν μπαίνει μπαίνει στα θεμέλια. Όχι, δεν συμφωνούμε. Για μας τα θεμέλια είναι η θεωρητική επιστήμη και οι περιφαριακοί πυλώνες είναι οι εφαρμοσμένες επιστήμες. Σε αυτό το foundation λοιπόν ε, ενσωματώνουμε τις γενικές αρχές και στους πυλώνες εφαρμόζουμε και το εφαρμόζουμε σε τρεις διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους, Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικό. Και εάν δούμε τις οικονομικές προκλήσεις, την ε, ειρήνη, τη σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή σε κάθε μία από τις τρεις γεωγραφικές περιοχές, η στόχευση, το ζήγεσμα, το σημείο εξισορρόπησης, οι προτεραιότητες, ο τρόπος επίτευξης όλων αυτών είναι διαφορετικά. Όμως πρέπει να, να ξεκινήσουμε με κάτι που το έχουμε από κοινού, το μοιραζόμαστε, δηλαδή τα θεμέλια. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η παράλληλη διαπραγμάτευση για αυτή την ε, στρατηγική δεν είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Είναι θεμελιώδης, ε, ζήτημα αυτό που θα συζητήσουμε. Όμως δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε ένα διαφορετικό, ξεχωριστό και παράλληλο σύμπαν. Με εκπλήσει το γεγονός ότι ακούσαμε τρεις Αφρικανούς πρέσβεις να παίρνουν το λόγο και βλέπουμε ότι υπάρχουν νέες απαντήσεις μεταξύ των διαφόρων θέσεων. Όλοι ελπίζουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να δούμε ότι συγκλίνουν οι απόψεις μεταξύ όλων μας. Και ερχόμαστε τώρα στη θεσμική δομή. συνδέονται αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι όλα ασπρόμαυρα ή άσπρα ή μαύρα. Η θεσμική δομή πρέπει να είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένη με τη δομή και τη διάρθρωση της συμφωνίας. Άρα να ενισχύουμε τις συνεδριάσεις μεταξύ Ευρωπαίων και Αφρικανών ομολόγων, μεταξύ Ευρωπαίων ομολόγων και ομολόγων της Καραϊβικής ή του Ειρηνικού. Όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα. Είτε σε υπουργικό επίπεδο, είτε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο στελεχών. Δεν σημαίνει ότι το ένα αποκλείει το άλλο. Αλλά να εφαρμόσουμε τη λογική ε, των θεωρητικών επιστημών και των εφαρμοσμένων επιστημών στη συμφωνία, τότε θα μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε. Και το πώς θα γίνουν όλα αυτά, αυτό θα είναι το προϊόν της διαπραγμάτευσης. Έχουμε τη δική μας άποψη, οι εταίροι μας έχουν τη δική τους άποψη, θα τα βρούμε κάπου αλλά αν συμφωνήσουμε όμως επί της προσέγγισης, ότι δηλαδή η θεσμική διάρθρωση της συμφωνίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο ε, ε διακύμεθα τη στάση μας εναντί αυτής της συμφωνίας. Και έρχομαι τώρα στην οικονομική στήριξη. Βεβαίως θα υπάρξει οικονομική στήριξη. Εμείς έχουμε υποβάλει τις ιδέες μας γίνονται διαπραγματεύσεις με τις αρχές τις υπεύθυνες για τον προϋπολογισμό Καθορίζουμε τώρα το χρονοδιάγραμμα με το Συμβούλιο, με την Αυστριακή Προεδρία και έχουμε κάποιες ενδείξεις για ε, το ύψος της χρηματοδότησης που προβλέπουμε για κάθε μία από τις περιφέρειες. Έρχομαι τώρα στην ουσία της συμφωνίας. Βλέπουμε τις αποκλήσεις, αλλά μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Τέλος, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Να ξεκινήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου και να προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και όσο πιο μακριά μπορούμε εντός ε, της ε, θητείας ε, των υφιστάμενων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή λειτουργεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά το Κοινοβούλιο θα έχει εκλογές λίγο νωρίτερα. Άρα ε, πρόθεσή μας είναι να κινηθούμε όσο το πιο γρήγορα για να καλύψουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση, αλλά είναι αδύνατο να δεσμευτούμε για κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να έχουμε διαφάνεια και θέλουμε και με την ομάδα εργασίας για το ΑΚΕ να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και με εδώ στην Επιτροπή σας να συνεργαστούμε με εσά για να γίνουν απολύτως κατανοητά τα ζητήματα και το πώς θα τα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και μα τελείωσε ο χρόνο. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκόμε και αν περισσέψει χρόνο, θα μπορείτε κι εσεί να ε, κάνετε κάποια συμπερασματικά σχόλια. Σα ευχαριστώ. Το κύριο ερώτημα είναι οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη και αν θέλουμε να παραμείνουν οριζόντιοι. Αυτό που είναι που ρώτησε η κυρία Χόιμπουχ. Πώς μπορούμε τώρα να δημιουργήσουμε μια διεθνή ε, δομή ε, στην οποία να για την οποία να συμφωνούμε όλοι. Χρειάζεται να, υπάρχουν... να υπάρχει πολυμερή συμφωνία, ε, όπως για παράδειγμα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Τα... Και για τη μετανάστευση ισχύει αυτό. Χρειάζεται μια παγκόσμια συμφωνία για την ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση. Αυτό υπάρχει και αυτό που μου μένει είναι εμείς να το αξιολογήσουμε και να το υποστηρίξουμε. Διότι η στήριξή μας θα επιτρέψει τη δημιουργία κοινών ε, δράσεων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Τώρα τα υπόλοιπα ζητήματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα, συνδέονται με πολλά, με τη φτώχεια πρώτον, με τη δομή της κοινωνίας και με ε, τη θέση που νομίζουν οι πολίτες πως έχουν σε αυτή. τα την αποξένωση της ε, νεολαίας, γι' αυτό και βλέπουμε να ε, στρατολογούνται νέοι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Και πρέπει λοιπόν να δούμε τις πραγματικότητες αυτές και να τις αντιμετωπίσουμε με μια ε, πολυμερή αντιμετώπιση. Επίσης, χρειάζεται να κινητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών, οι οργανώσεις πολιτών και να δούμε τι είδους επενδύσεις θέλουμε να κάνουμε. Επενδύσεις οι οποίες θα ε, βοηθούν και δεν θα ε, καταλυστεύουν τις περιοχές αυτές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές, στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Θεωρώ όμως ότι το ζήτημα της μετανάστευσης, παρά τον πολύπλοκο χαρακτήρα του, δεν σημαίνει ότι είναι και δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ε, πρέπει να δούμε το γενικότερο πλαίσιο, ποιος επωφελείται από αυτό, ε, πού πηγαίνουν οι ροές, όχι μόνο ε, να στεκόμαστε στην βοήθεια την οικονομική, να δημιουργούμε ταμεία κτλ, να δούμε το γενικότερο πλαίσιο. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, μέσα στην ε, Κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο οι υποεπιτροπές οι οποίες ε, θα συζητούν τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αρκεί μόνο να συναντιόμαστε μια φορά στο τόσο και να συζητούμε, αλλά να υπάρχει ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα δράσης για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ε, αυτά. Και νομίζω πως έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Θα σταματήσω όμως εδώ και θα σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Κρίστιαν, ένα λεπτό για τα τελευταία λόγια. Καταλαβαίνω αν οι διερμηνείς θέλουν να φύγουν. Um, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Συμφωνώ απόλυτα με όσα λέτε. Κύριε Γκόμεζ, να σας ε, Υπενθυμίσω ότι γίνεται λόγος για πυλώνες, για θεμέλια. Οι πυλώνες δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους αν δεν υπάρχουν γερά θεμέλια και εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση. Αλλά να αναγνωρίσουμε και τις αλλαγές που έχουν γίνει. Μην ξεχνάτε ότι όταν υπεγράφει η Συμφωνία του Κοτονού δεν υπήρχε Αφρικανική Ένωση. Υπήρχαν άλλες τομές. Υπήρχε ε, επίσης ε, μεν το φόρουμ των νήσων του Ειρηνικού, αλλά είχε μόλις συσταθεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πραγματικότητα είναι διαφορετική, τα επίπεδα ανάπτυξης και φιλοδοξίας διαφέρουν επίσης και αυτό πρέπει να το ε, αναγνωρίσουμε και να αντικατοπτρίζεται στην πολιτική μας και στους κοινού πυλώνες, τα κοινά θεμέλια. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είπα και τόνισε και η κυρία Χόιμπουχ και η κυρία Ρένα, έχουν ένα κεντρικό πλαίσιο. Και ε, αυτό καλύπτει όλους τους τομείς πολιτικής. Η τομή πολιτικής όμως που ανέφερε η κυρία Χιμένες, για παράδειγμα, διακυβέρνηση, ασφάλεια, άμυνα, μετανάστευση, όλα αυτά είναι διαφορετικού μεγέθους προκλήσεις ε, για παράδειγμα, για τις χώρες του Ειρηνικού, από ό,τι για την Αφρική. Και θα ήταν ανόητο να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσει. Γι' αυτό χρειάζεται